Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην ακρόαση αυτή για τους προτινόμενους κανόνες όσον αφορά το σεβασμό του ιδιωτικού βίου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας καλωσορίζω όλους και τους φιλοξενούμενους μας βέβαια. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και σημαντική υπόθεση η η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή μας από τη ΛΥΜΠΕ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή Μαριλόστεν και τους σκιώδες συγητές για την υπόθεση αυτή που είναι εδώ παρόντες. Έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά για αυτό το τόσο σημαντικό φάκελο. Στη σημερινή ακρόαση έχουμε μαζί μας πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Θα μας παρουσιάσουν το πλαίσιο λοιπόν του θέματος που μας απασχολεί και ελπίζω ότι θα έρθουν όλο και περισσότεροι ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Θα σας παρουσιάσω καταρχήν λιγάκι εγώ το πλαίσιο τι συζητάμε σήμερα και μετά θα περάσουμε στην παρουσίαση των τριών πάνελ που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο πάνελ θα μιλήσουμε για τα θεσμικά ζητήματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η ακρόαση αυτή καταρχήν να ξέρετε ότι μεταδίδεται από το διαδίκτυο και όλε, οι παρεμβάσει των ομιλητών και των συμμετοχών, θα μαγνητοσκοπούνται. Γιατί πράγμα συζητάμε λοιπόν. Συζητάμε για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υποβλήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2017 πρόταση κανονισμού για την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που ονομάζεται e-Privacy Regulation και ακολουθεί την αντίστοιχη οδηγία που είχαμε το 2002 η οποία φροντίζει για τους κανόνες που προστατεύουν τον ιδιωτικό βίο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμπληρώνει επίσης και κάνει πιο συγκεκριμένη την Οδηγία 9546 για την προστασία των δεδομένων. Θέλει λοιπόν να προστατεύσει το απόρριτο των επικοινωνιών να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα μάλιστα και με το άρθρο 7 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προτινόμενος κανονισμός λοιπόν λαμβάνει υπόψη τώρα τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις οικονομικές εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Υπάρχουν νέες υπηρεσίες που υπάρχουν παράλληλα με άλλες πιο παραδοσιακές επικοινωνίες που είχαμε κατά το παρελθόν. Αλλά πρέπει να καλύπτονται εξίσου και η ΜΕΝ και η ιδέα από τους κανόνες προστασίας του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων. Μέχρι τώρα όμως δεν υπήρχε αυτή η προστασία και για τις δύο περιπτώσεις από την Οδηγία 2002 58. Ο προτινόμενος κανονισμός λοιπόν ενημερώνει κατά κάποιο τρόπο την οδηγία αυτή και την ευθυγραμμίζει με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία έχουμε και από τον Γενικό Κανόνα για την Προστασία των Δεδομένων. Έτσι λοιπόν τώρα προβλέπεται κάλυψη και των νέων μορφών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να υπάρχει το ίδιο επίπεδο προστασίας των ε, ατόμων ανεξάρτητα από το ποιο είδος ηλεκτρονικών επικοινωνιών χρησιμοποιούν λαμβάνει υπόψη την εμπειρία που έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια με τα cookies και ό,τι άλλο καινούριο έχει μπει στην ζωή μας σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι κανόνες του κανονισμού αυτού δεν πρέπει να μειώσουν ε, βέβαια το επίπεδο προστασίας βάσει του κανονισμού για την ε, προστασία δεδομένων. Η σημερινή πρόταση συνεισφέρει και για να Επιτευθεί η στρατηγική μας για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αντιμετωπίζονται εδώ τα διάφορα θέματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ακρόαση αυτή και γι' αυτό συμμετέχουν στην ακρόασή μας διάφοροι τομείς, τηλεπικοινωνίες, νέες υπηρεσίες παρόχων επικοινωνιών, οι καταναλωτές με κυβερνητικές οργανώσεις, καθηγητές, αρχές προστασίας δεδομένων κλπ. Έχουμε ένα καταπληκτικό πάνελ ομιλητών που σίγουρα θα συμπληρώσουν την εισαγωγή μου αυτή και θα μας βοηθήσουν σε βάθος να εξετάσουμε το θέμα μας. Μετά τις παρουσιάσεις θα έχουμε και ερωτήσεις και απαντήσεις. Πείτε εδώ στο συνάδελφο αν θέλετε να πάρετε το λόγο μετά τους προσκεκλημένους μας όσο κάνουν τις παρουσιάσεις τους, δηλαδή προσκεκλημένοι μας, ενημερώστε τη γραμματεία αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Λοιπόν, σε αυτό το πρώτο τμήμα θα ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε την παρουσίαση της κυρίας Δέσποινα Σπανού, που είναι Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Connect. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράης. Όντω έχετε καταφέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Βλέπω τόσο πολύ κόσμο εδώ, παρόλο που είναι μια εβδομάδα που συνήθως ο κόσμος παίρνει διακοπές. Το ότι είναι εδώ λοιπόν παρόντε τόσοι ευρωβουλευτές και τόσος κόσμος είναι μεγάλη τιμή για μας. Και δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόταση. Πρόσφατα εδώ και λίγους μήνες ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Πριν ήμουνα στους καταναλωτές Κάποιοι από εσά το γνωρίζετε αυτό ήδη. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν ασχολιόμουν με τους καταναλωτές είδαμε εκεί να υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που ασχολιόταν με την προστασία των καταναλωτών στις επικοινωνίες ακριβώς. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές, αλλά συγχρόνως θέλουν να προστατεύονται τα δικαιώματά τους και ο ιδιωτικό τους βίος. Και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρόσφατη εξέλιξη της Παρασκευής, όταν οι υπουργοί του G20 συμφώνησαν στη δήλωσή τους για την ψηφιακή οικονομία να λάβουν υπόψη τους και θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών. Και αυτό βασιζόμενοι σε μια διάσκεψη που έλαβε χώρα τον προηγούμενο μήνα για την προστασία των δεδομένων και κυρίως του ιδιωτικού βίου. Ήταν ένας από τους δέκα πιο σημαντικούς τομείς, τους οποίους πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάθε φορά που μιλάμε για την ψηφιακή ε, μεταλλαγή της κοινωνίας μας. Θέλω επίσης να πω ότι στη διάσκεψη αυτή η Ευρώπη ε, θεωρήθηκε ως ε, έχοντα ηγετικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, όχι μόνο γιατί έχουμε κανόνες για αυτό το θέμα που άλλοι δεν έχουν, αλλά γιατί έχουμε και σύγχρονους κανόνες. Στο λίγο χρόνο λοιπόν που έχω στη διάθεσή μου θα σας εξηγήσω τη λογική πίσω από την πρόταση. Πρώτα απ' όλα γιατί προτείναμε κάτι για την προστασία ε, στις ε, ηλεκτρονικές επικοινωνίες του ιδιωτικού βίου. Και μετά ευχαριστώ να συζητήσουμε μαζί περισσότερο. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος, ο προφανής, είναι η ίδια προστασία του ιδιωτικού βίου. Ό,τι γράφει, λέει προφορικά στις επικοινωνίες του κανείς πρέπει να προστατεύεται. Όταν ε, είχαμε αλληλογραφία με γράμματα, τα κρατούσαμε για τον εαυτό μας. Τώρα, με την κυκλοφορία των δεδομένων, την ηλεκτρονική, αλλάζουν τα δεδομένα και πρέπει να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε τα συμφέροντα του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τις αποφάσεις του. Ο δεύτερος λόγος είναι να μην ε, προστατεύουμε μόνο τους ανθρώπους, τα ε, φυσικά πρόσωπα, αλλά να προστατεύουμε και τα νομικά πρόσωπα. Δεν πρόκειται μόνο δηλαδή για το γενικό κανόνα που αφορούσε τα φυσικά άτομα. Εδώ πέρα μιλάμε και για νομικά πρόσωπα, διαφορούς κλάδους τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις κτλ. που φυσικά και έχουν και αυτοί απόρριτα. Και ο τρίτος λόγος για την Ευρώπη ήταν ότι πρόκειται εδώ πέρα και για την ελευθερία του λόγου, αλλά και για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πληροφορίες πρέπει να διαχέονται όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των ε, επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν θελήσαμε να έχουμε έναν κανονισμό εξυγχρονίζοντας ε, όλους αυτούς τους τομείς. Βέβαια, το εύρος εφαρμογής του κανονισμού είναι διαφορετικό από εκείνο των οδηγιών. Πρόκειται για το άρθρο 8 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η πρόταση αυτή αποτελεί την ερμηνεία του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία των απόρριτων επικοινωνιών όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7. Το έβρος εφαρμογής λοιπόν είναι διαφορετικό πρέπει να επεκτείνουμε συνεπώς την προστασία των δεδομένων όχι μόνο στα πρόσωπα και στα νομικά πρόσωπα, αλλά να φροντίσουμε ότι καλύπτεται το απόρριτο, ότι προστατεύεται. Ποιοι είναι οι στόχοι τώρα τη πρόταση αυτή. Πρώτος στόχος είναι υψηλό επίπεδο προστασίας για να ισχύουν κανόνες που προστατεύουν πραγματικά πολύ τις ε, ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο κύριος Μωράης πριν από λίγο είπε ότι ο στόχος της πρότασης είναι να λάβει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι έχουμε νέου είδους υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι πολίτες, οι καταναλωτές μας. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει μια συνένεση στους κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες μας και που να ισχύουν και στα τρίτα μέρη. Οποιοδήποτε δηλαδή χρησιμοποιεί ε, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή θέλει να ε, αποθηκεύσει δεδομένα ή θέλει να χρησιμοποιήσει cookies ή οτιδήποτε. Όλα αυτά βέβαια αντικατοπτρίζουν έργο που έχει ήδη γίνει. Για τα cookies για παράδειγμα. Υπάρχει ε, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που ήδη από το 2015 ασχολείται και είπε ότι πάνω από 16.000 cookies υπάρχουν σε διάφορες ιστοσελίδες. Το νούμερο είναι τεράστιο. Με ημερομηνία λήξης πολύ αργά και θέλουμε να δούμε πώς, με ποιο τρόπο πετυχαίνει τη συνένεση εκείνου ο οποίος επικοινωνεί. Δηλαδή, ο καταναλωτής είναι όντως ενήμερος για το ότι δίνει τη συγκατάθεσή του με τα κούκκι σε διάφορες να παρακολουθούν το τι κάνει. Πώς θα γίνει αυτό. Πρώτον, οι browsers να εμποδίζουν τρίτα μέρη να αποθηκεύουν πληροφορίες και ο δεύτερος τρόπος είναι οι browsers αυτοί, οι φιλομετρητές, να μπορούν εύκολα να επιλέξουν τις ρυθμίσεις προστασίας, ιδιωτικότητας που έχει επιλέξει ο καθένας. Να γίνεται αυτό με επιτυχία δηλαδή. Ο δεύτερος στόχος ήταν να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες. Ήταν πολύ σημαντικό όλοι όσοι προσφέρουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην αγορά να υποβάλλονται στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο χωρίς να εμποδίσεται η καινοτομία. Θέλουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει νομική βεβαιότητα ένα νομικό πλαίσιο, αλλά να μπορεί να εισαχθεί η τεχνολογία, καινοτομίε, οτιδήποτε νέο έρχεται. Κάποιοι χρησιμοποιούν για συγκεκριμένους λόγους το διαδίκτυο και μόνο. Οι πάροχοι λοιπόν πρέπει να μπορούν να συνάδουν και με τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες, αλλά να δεσμεύονται κιόλα. Ο τρίτος στόχος ήταν να διασφαλίσουμε συνοχή με, τους, με τις ρυθμίσεις για την προστασία δεδομένων που έχουμε υιοθετήσει μέχρι τώρα και με τα κριτήρια που έχουν αποφασίσει οι νομοθέτες. Συνεπώς θέλουμε συνοχή και για τους ορισμούς αλλά και για την κάλυψη. Υπάρχει όμως και ένας τέταρτος στόχος που δεν πρέπει να ξεχνάμε για το πρόβλημα με όλους αυτούς τους κανόνες είναι το πώς εφαρμόζονται. Στην πρόταση αυτή λοιπόν έχουμε ευθυγραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες γιατί θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται από τις ίδιες αρχές που θα έχουν τη γνώση, την πρόσβαση στην αγορά και θα φροντίζουμε τον ίδιο τρόπο και με συνοχή να εφαρμόζονται οι κανόνες. Αυτή λοιπόν ήταν η στόχη μας. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε ήδη συζητήσει σε επίπεδο ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση υπό Μαλτέζικη Προεδρία. Και ελπίζουμε μετά να μπορέσουμε πιο γρήγορα η Προεδρία να προχωρήσουμε. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντοπίζουμε έτσι τους τομείς πάνω στους οποίους θα χρειαστεί παρετέρω συζήτηση. Και ελπίζω η σημερινή συνάντηση να προσφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσματα και να μας τροφοδοτήσει με καλές νέες ιδέες. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε γνωμοδότηση από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που καλωσορίζει την πρόταση αλλά εντοπίζει και όλες κάποιες αδυναμίες αυτήν. Όσον αφορά το επίπεδο προστασίας, λένε ότι δεν είναι αρκετά υψηλό. Μετά τις πασχαλινές διακοπές περιμένουμε τις αρχές του επόπτη προσωπικών δεδομένων να μας δώσει τη δικιά του γνωμοδότηση. Το πιο σημαντικό πάντως για τις αγορές, για τις αρχές και για τους πολίτες πιστεύω ότι είναι να εγκριθεί ο κανονισμός όσο γίνεται πιο γρήγορα με την εφαρμογή του Γενικού Κανόνα που είναι το Μάιο του 2019 για να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση. Ευχαριστώ και νομίζω δεν ξεπέρασα το χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ Βέσπινα. Αυτό μας αφήνει και χρόνο για τις ρωτήσεις που είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι τώρα θα ακούσουμε, θα έχουμε μάλλον την γνωμοδότηση του Επόπτη Προστασία των Δεδομένων ε, το Μάιο, αλλά ο κύριος Μπουταρέλη είναι εδώ σήμερα, ε, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασία των Δεδομένων και θα θέλαμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα σας πω ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια ε, πρώτερη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την ευγενική σας πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με μια προσωπική ιστορία, καθώς ε, αισθάνομαι ότι είμαι προσωπικά κοντά σε σχέση με το θέμα της ιδιωτικότητας, ε, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ε, πριν λίγα χρόνια ήμουν ο εκπρόσωπος της Ιταλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, της ε, προστασίας της ιδιωτικότητας ό,τι αφορά τμήμα του κανονισμού του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ε, μιλώ για την οδηγία 9766. Τότε συζητούσαμε την συμπλήρωση γενικών διατάξεων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων οριζόντια. Και 20 χρόνια μετά προσεγγίζουμε ένα νέο κεφάλαιο αυτή τη φορά έναν κανονισμό που στοχεύει στο να ε, συμπληρώσει και να διευκρινίσει γενικές διατάξεις στο γενικό κανονισμό και πάνω κάτω έχουμε τα ίδια ζητήματα σε ό,τι αφορά την ε, συνάφεια όπως υπόθηκε, ε, σε ό,τι αφορά τη συνεκτικότητα, σε ό,τι αφορά το να μην μειώσουμε τις υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με το να είμαστε επιλεκτικοί, να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι και να προσανατολιζόμαστε και προς το μέλλον. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι πολύ που θα σας παρουσιάσω σήμερα την εμπειρία μου, αλλά και κάποιες σκέψεις για την πρόταση. Με αυτόν τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής της ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ένα πλαίσιο προστασίας των δεδομένων σίγουρα δεν θα ήταν ολοκληρωμένο. Ο κανονισμός προστασία των δεδομένων σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτή τη θητεία. Όμω ε, χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο νομικό εργαλείο για να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, όπω το εγγυάται το άρθρο 7 τη χάρτα. Και όπως είπαν και τα δύο δικαστήρια για το άρθρο, η εμπιστευτικότητα, το απόρριτο των πληροφοριών είναι ουσιώδες συστατικό. Έτσι λοιπόν, όπως είδαμε και στην πρόσφατη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας ε, του Άρθρου το 29, εγώ καλωσορίζω και υποστηρίζω την Κομισιόν που θέλει να κάνει ακριβώς αυτό. Επίσης, υποστηρίζω την επιλογή του νομικού μέσου, δηλαδή ενός κανονισμού, που όπως γνωρίζετε, όχι μόνο θα εφαρμοστεί άμεσα, αλλά μπορεί και να συνεισφέρει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο εναρμόνισης και συνεκτικότητας. Και τέλος, Καλωσορίζουμε τη φιλοδοξία της πρότασης να παρασχεί ένα υψηλότερο και καλύτερο επίπεδο προστασίας ως προς το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα. Αν αυτό είναι ο στόχος, υποστηρίζουμε πλήρως την ιδέα του να καταστήσουμε τις υποχρεώσεις απορρίτου εφαρμόσιμες σε ένα ευρύτερο σε μια ευρύτερη γκάμα παρόχων και υπηρεσιών και στις επιφύσεις υπηρεσίες, over the top services, που αντικατοπτρίζουν την πρόοδο των τεχνολογιών και τις ε, αλλαγές ε, στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε. Σήμερα χρησιμοποιούμε όλα και περισσότερες εφαρμογές και συνδεδεμένες συσκευές σε σύγκριση με κάποια χρόνια πριν. Αναφέροντας και άλλα θετικά στοιχεία, όπως έκανε και η ομάδα εργασία του έρθρου 29 την περασμένη εβδομάδα, θεωρούμε και εμεί ότι η πρόταση χορήγηση ε, αρμοδιότητας επιβολή ε, στι αρχέ προστασία των δεδομένων, ε, κυρίω σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα του μηχανισμού συνάφεια εντό του Συμβουλίου τη προστασία των Δεδομένων θα συνεισφέρει σε πιο αποτελεσματική επιβολή των κανόνων περί απορρίτου υπό το νέο κανονισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε την περσμένη εβδομάδα η ομάδα εργασία του άρθρου 29, έχουμε κάποιε ανησυχίε. Σε σχέση με τον η πρόταση ω έχει, μπορεί πράγματι να υλοποιήσει την υπόσχεσή τη, δηλαδή να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασία τη ιδιωτική ζωή τη ηλεκτρονική επικοινωνία. Γιατί το κάνουμε αυτό, Καταρχήν, λόγω τη πολυπλοκότητα των προτινόμενων κανόνων, οι επικοινωνίε όλο ένα και περισσότερο ε, χρησιμοποιούν με τα δεδομένα, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα που στέλνονται από τερματικό εξοπλισμό και όλα αυτά χρήζουν διαφορετικού επίπεδου απορρίτου και αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί ξαφνικά να παρουσιάσει ένα κίνδυνο ε, κάποιων κενών μη στην προστασία. Δεύτερον, να πω ότι οι περισσότεροι από τους ορισμούς επί των οποίων βασίζεται η πρόταση θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση και απόφαση σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, στο πλαίσιο ενό διαφορετικού νομικού μέσου του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνιών. Δεν υπάρχει νομική αιτιολόγηση σήμερα για σύνδεση των ε, δύο μέσων τόσο στενά και οι ορισμοί του ανταγωνισμού και που επικεντρώνονται στην αγορά του κώδικα δεν είναι κατάλληλοι για το σκοπό στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επομένως, στην γνωμοδότηση που θέλουμε να δημοσιεύσουμε, αμέσως μετά το Πάσχα, θέλουμε να ζητήσουμε τη συμπερίληψη ενός συνόλου απαραίτητων ορισμών στον κανονισμό e-privacy, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους στόχους και το πεδίο εφαρμογή. Τρίτον, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από υπεύθυνου τη επεξεργασία άλλου από του παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που καλύπτονται την πρόταση αυτή. Η πρόσθετη λοιπόν προστασία που προσφέρεται στα δεδομένα τηλεπικοινωνιών δεν θα έχει νόημα αν μπορούσε να καταστρατηγηθεί εύκολα, παραδείγματο χάρη με τη μεταφορά των δεδομένων σε τρίτα μέρη. Το επίπεδο της προστασία θα πρέπει να εξαρτηθεί στην ευαίσθητη φύση της πληροφορίας και όχι στο ποιος είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο αρμόδιος της επεξεργασίας. Τέλος να πω ότι δεν θα πετύχουμε τη φιλοδοξία να προστατεύσουμε το απόρριτο των επικοινωνιών χωρίς ισχυρές απαιτήσει ε, για σχεδιασμό εξορισμού και εξχεδιασμού που τουλάχιστον θα πρέπει να συμβαδίζουν με αυτά που υπάρχουν στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Πολλοί συμφωνούν με αυτές τις ανησυχίες ε, στην ε, ομάδα εργασία στο άρθρο 29. Το βλέπουμε αυτό και στην τελευταία γνωμοδότηση, αλλά και στην γνωμοδότηση 1-2017 που υιοθετήθηκε στις 4 Απριλίου. Και εγώ συνεισέφερα σε αυτή ως μέλος της ομάδας εργασίας. Κατά τη γνώμη μας, Στη γνωμοδότησή μας, με συγχωρείτε, θα κάνουμε προτάσεις για το πώ να λύσουμε τα πλέον πιεστικά θέματα με πλήρη συνεργασία με τη γνωμοδότηση της ομάδας του άρθρου 29, επικεντρωνόμενη σε τομεί όπου υπάρχουν σοβαρότερες ανησυχίες, άλλους ε, τομεί όπου έχουμε και λοιπέ ανησυχίες, αλλά και κάποιες λεπτομέρειες που χρήζουν αποσαφήνισης στοχεύουμε συγκεκριμένα στο να δώσουμε μια, πρόσφα... μια πρόσθετη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τα πιο ευαίσθητα θέματα, όπως πούμε το σχάρι, τους ε, τείχους κούκι, τους cookie walls και ε, το νομικό ε, δυναμική αιτιολογία του νόμιμου συμφέροντος, ε, όπως εφαρμόζεται στα μεταδεδομένα. Επίσης, ε, να δούμε τι ισχύει σε ό,τι αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σε τομείς πέρα από την επιβολή του δικαίου. Για να πάω τώρα πέρα από το θέμα του στόχου είναι να συμπληρωθούν και να διευκρινιστούν οι φυστάμενες διατάξεις στο γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Τι σημαίνουν αυτά κατά τη δική μου γνώμη, ότι υπάρχει μικρή δυνατότητα για προσαρμογές. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πλήρη συνεκτικότητα και συνέπεια. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιλεκτικοί. Επί της αρχής σημαίνει πλήρη υποστήριξη να αυξήσουμε τις υφιστάμενες ασφαλιστικές δικλίδες και όχι να μειώσουμε όσα διαπραγματευτήκαμε ήδη πριν τέσσερα χρόνια και σε αυτό το κοινοβούλιο. Επίσης, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μελλοντικό νομικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλου του φορεί, σε όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματο ε, θα μεταφερθούν στο πλαίσιο εκείνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν ε, προσέφερα τα 15 ε, δευτερόλεπτα, αλλά τέλος πάντων σεβάστηκα το χρόνο. Ευχαριστώ. Γιατί όλοι αναφέρουν το χρόνο. Έχω τόσο κακή φήμη ότι σας πιέζω να σέβεστε το χρόνο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ο τρίτος μας ομιλητής είναι ο κύριος ε, Μπορκίσιος, ο οποίος θα παρουσιάσει τα ε, προκαταρκτικά αποτελέσματα της ε, μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικέ επικοινωνίες που ανατέθηκε από το θεματικό τμήμα δικαιωμάτων των πολιτών και συνταγματικών υποθέσεων. Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, έχει διάφορα ενδιαφέροντα όπως είναι ε, διάφορα ενδιαφέροντα. Έχετε το ε, λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκπροσωπώ την ομάδα που έγραψε την συγκεκριμένη πρόταση. Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ ε, για τη συγκεκριμένη πρόταση, όμως επειδή έχουμε μόνο 10 λεπτά ε, θα ε, αναφερθώ στα τέσσερα πιο αδύναμα σημεία. Τέσσερα σημεία λοιπόν, αφενός ο εντοπισμός του Wi-Fi, η εξορισμού προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα tracking walls και η εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών. Αρχικά λοιπόν όσον αφορά τον εντοπισμό του Wi-Fi, ε, που διαβάζοντας ε, το άρθρο 8 ορίζει ε, η παρακολούθηση ανθρώπων στους δρόμους παρακολουθώντας το σήμα του Wi-Fi επιτρέπεται χωρίς την έγκρισή του σε περίπτωση που η εταιρεία δηλώσει ότι αν πεπατάτε έξω τότε ε, μπορούμε να σας εντοπίσουμε. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Το πόστρο λοιπόν θα πρέπει να λέει το πώς οι άνθρωποι θα μπορούν να περιορίσουν αυτή την ε, παρακολούθηση όπως για παράδειγμα να λέει απενεργοποιήστε το κινητό σας ή το wifi σας. Δεν νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε ε, έναν κανόνα δύο μερών, ο οποίος θα είναι καλύτερος σε αυτόν, ο οποίος θα ορίζει ότι ε, η παρακολούθηση του Wi-Fi θα επιτρέπεται μονάχα ύστερα από ενημερωμένη έγκριση από ε, τον εκάστοτε χρήστη και δεύτερον, σε περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα cloud μέσα στην πόλη, τότε θα μπορούμε να υπολογίσουμε τα πλήθη, όμως ε, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διασπαρμένα και ανώνυμα, ε, να δούμε δηλαδή σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση και πού όχι, χωρίς όμως η εταιρεία να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί με μονομένους χρήστες. Ε, το άρθρο 29 δίνει προτάσεις για δυνατότητες ασφάλειας. Το επόμενο θέμα τώρα το οποίο είναι εύκολο ε, θέμα. Η ε, πρόταση ε, στο άρθρο 10 ορίζει ότι οι φιλομετρητές θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες σχετικά με την παρακολούθηση. Η αρχική εκδοχή που θεωρούμε ότι είναι καλύτερη είναι ότι θα πρέπει οι φιλομετρητές να έχουν φιλική και ρυθμίσεις ε, προς τους ε, χρήστες ε, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Την προηγούμενη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λοιπόν στην ομάδα εργασίας επιθυμούμε να έχουμε μια πιο ουδέτερη τεχνολογικά ταυτότητα η οποία θα εξετάζει τον κανονισμό του e-privacy που θα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείε tracking να, να τηρούν πρότυπα do track διότι αυτά δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να πούν όχι σε ό,τι αφορά τα cookies ε, και τα λοιπά. Συνολικά λοιπόν οι φιλομητρές θα πρέπει να έχουν ε, τέτοιες δυνατότητες εύκολες προς το χρήστη. Και τέλος έχουμε τα, στη συνέχεια έχουμε τα ε, tracking walls, ε, οι cookie walls, ε, τύχη cookie, εδώ έχουμε μια, ε, ένα δημοφιλές μήνυμα, ένα σύνηθες μήνυμα που εμφανίζεται, μπαίνετε σε μια ιστοσελίδα και πετάγεται αυτό το pop-up το οποίο λέει πατήστε στο πορτοκαλί κουμπί αν συμφωνείτε εμείς ε, και καμιά δεκαριά άλλες εταιρείες διαφημίσεων αλλά και εταιρείες ε, tracking θα μπορούν, αν συμφωνείτε λοιπόν, ε, να, ε, αν συμφωνείτε να δεχτείτε όλα αυτά τα ε, tracking cookies. Σε περίπτωση που πατήθετε όχι, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα. Γελιοποιεί λοιπόν την την έγκριση που δίνεται ε, με ελεύθερη βούληση. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Πάμε στην επόμενη διαφένεια Προ, ε, προτείνω δύο δυνατότητες. Αφενός ε, μπορούμε απλά να απαγορεύσουμε αυτά τα τείχη τα οποία θα ήταν και η πιο εύκολη λύση με έναν απλό ξεκαθαρό κανόνα. Όμως μπορούμε να έχουμε μια, πιο, μια διαφορετική προσέγγιση και να ορίσουμε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες τέτοια τείχη δεν θα επιτρέπονται θα μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό με τις ε, ε, γκρι και μαύρες λίστες. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, ε, θα μπορούμε να έχουμε ιστοσελίδες του δημόσιου τομέα, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν τέτοια τύχη ή και άλλες ιστοσελίδες με ευαίσθητα δεδομένα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοια τύχη σελίδες που έχουν ε, θέση ε, που μοιάζει με μονοπόλιο. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν τέτοια τύχη. Ε, είναι πιο πολύπλοκο αυτό, όμως είναι πιο ξεκάθαρο, το οποίο υποστηρίζει την, σε αντίθεση με την πρώτη εναλλακτική που προβλέπει μια πλήρη απαγόρευση. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Το τέταρτο και τελευταίο θέμα αφορά το απόρτο των επικοινωνιών. Πολύ ε, γενικά το άρθρο 5 και 6 ορίζει ότι υπάρχει απαγόρευση της παρακολούθησης ε, των επικοινωνιών, ε, δεν θα πρέπει να παρακολουθούνται τηλεφωνήματα και email σε περίπτωση που υπάρχει μια εξαίρεση, όπως είναι για παράδειγμα για λόγους ασφαλείας του δικτύου ή εάν υπάρχει η συνένεση του χρήστη. Συνολικά λοιπόν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα καλό σύστημα για να ρυθμιστεί όλο αυτό. Όμως το σύστημα μπορεί να βελτιωθεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όλοι οι χρήστες ε, θα πρέπει ε, να εγκρίνουν την ανάλυση των για την ανάλυση των ε, επικοινωνιών τους ε, δεν γίνεται να υπάρχει κάποιος πάροχος ο οποίος κάνει ε, εξόρυξη δεδομένων. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε εγκρίνει κάτι τέτοιο, γι' αυτό το λόγο όλοι οι χρήστες θα πρέπει να το εγκρίνουν σε παρέμβαση των επικοινωνιών τους, κάτι το οποίο είναι πασιφανές βέβαια. Και φυσικά υπάρχουν, ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων, όπως είναι για παράδειγμα για την ασφάλεια ε, του δικτύου, για, την, ε, για το φιλτράρισμα από ε, SMAM. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες, κάποιοι κανονισμοί για αυτό, όμως εμείς είμαστε κατά του να υπάρξει μια ανοιχτή εξαίρεση. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε θα είναι για παράδειγμα Ε, μέσω ε, ε, κανονισμών να δοθεί δυνατότητα να υπάρχουν εξαιρέσει. Φανταστείτε λοιπόν σε πέντε χρόνια να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η νέα τεχνολογία ε, έχει ε, εισαχθεί στη ζωή μας ε, με, όπου χρειάζεται νέα ανάλυση μεταδεδομένων και νέα τύχη και δεν προσκρούει σε κάποιους από τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα να προσθεθεί μια εξαίρεση και να επιλύσουμε το πρόβλημα του να σκεφτόμαστε σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχαμε προβλεφθεί. Ένα τελευταίο σημείο ε, το οποίο ε, προκαλεί και τις μεγαλύτερες διαφωνίες. Ε, η πρόταση ορθά προτείνει ότι οι πάροχοι επικοινωνιών θα πρέπει να παρέχουν το πορτό των επικοινωνιών. Συμφωνούμε απόλυτα. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι πασφανές. Όμως, μπορούμε να αναλογιστούμε και ε, ζητήματα σχετικά με την πιο αυστηρή ε, την αυστηροποίηση των ε, κανόνων, διότι οι πάροχοι μπορούν να εξετάσουν πολύ περισσότερο και να παρακολουθήσουν πολύ περισσότερο εκτός από το Skype ή το WhatsApp ή το Gmail αυτό το, ε, το οποίο αποκρυπτογραφούμε δεν μπορούν να το δουν, όμως το κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει πιο αυστηρούς τους κανόνες για τους παρόχους. Ε, έτσι λοιπόν, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρχει ε, η έγκριση από τους χρήστες, δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δυνατότητα στοχευμένου marketing, για παράδειγμα, από εταιρείε, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ένα ακόμα σχόλιο το οποίο θα πρέπει να είναι εμφανές, αλλά θα ήθελα να το σημειώσω, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε διαφορετικούς κανόνες e-privacy, παρόλο ε, που υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να χειροκροτήσετε, άφοβα. Είχα σταματήσει χειροκρότημα σε μια άλλη ακρόαση, αλλά είχα κάθε δικαίωμα σε αυτό. Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας και τώρα έχουμε αρκετό χρόνο για ε, ερωτήσεις. Γι' αυτό θα σας παρακολούσα να ε, περιοριστείτε στο χρόνο σας για να συζητήσουμε αρκετά. Θα ξεκινήσουμε ε, με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Με την Λόριστιν λοιπόν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους μας. Χωρίς τη δικιά σας συνεισφορά, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήδη μας βοηθάει με πολύ καλή συνεργασία και μια πολύ καλή πρόταση. Είναι μια πρόταση που μας εμπνέει να την βελτιώσουμε και όχι να αντιταθούμε σε αυτήν. Άρα είναι μια πολύ θετική κατάσταση αυτή. Θέλω όμως να ρωτήσω την Επιτροπή ακόμα. Σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε άτυπα, έτσι από διάφορες πηγές, φαίνεται ότι υπάρχει και μια πιο αυστηρή εκδοχή της πρότασης. Εδώ αναφέρεται για παράδειγμα η δυνατότητα να έχουμε εξορισμού προστασία του ιδιωτικού βίου από τους browsers βάσει των ρυθμίσεων. Ποιος όμως είναι ο λόγος που δεν έχουμε ακριβώς αυτή τη ριζοσπαστική μέθοδο που πολλοί θεωρούν ότι είναι μια θετική λύση. Επίσης, στα πανεπιστήμια θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Μπορούμε να έχουμε περισσότερα δεδομένα από τις δικές σας μελέτες. Μπορούμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την μελέτη σας αυτή. Όσο περισσότερα δεδομένα μπορείτε να μας δώσετε από τη μελέτη σας, τόσο το καλύτερο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι σκιώδεις εισηγητές. Τώρα, παρακαλώ, ο κύριος Πότη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, για την ακρόαση αυτή πρώτα απ' όλα και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις τους και αποτελούν μια πολύ καλή εισαγωγή για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την προστασία του ιδιωτικού βέλιου. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κανονισμό και φυσικά και θα πρέπει να είναι συμβατός με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ακούσαμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει κάποια σύνδεση και με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δεν είναι σαφέ όμω τι ορισμού χρειαζόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτησή μου. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε και να συζητήσουμε τελικά αλλαγέ ορισμών στι ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δεύτερον, μετά την παρουσίαση του κύριου Μπεργκέζο. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο ευθύ εξ αρχής να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε κάποια ισορροπία, κοιτώντας προς το μέλλον. Δεν ξέρουμε τι δυνατότητες θα έχουμε στο μέλλον. Η κατεξουδότηση πράξη αναφέρει εξαιρέσεις. Νομίζω έτσι θα είναι πιο εύκολο να συζητήσουμε γενικά τον κανονισμό Απ' την άλλη αυτά που είπατε για το, σημείο, για το άρθρο 8 σημείο 2 που έχει να κάνει με το Wi-Fi και αυτούς τους τείχους παρακολούθησης όπως λέγονται είναι σωστά. Θέλω να αναφερθώ και στα τρίτα μέρη. Τι συνέπειες απρόβλεπτες μπορεί να έχει μια τέτοια ρύθμιση στις τοπικές εφημερίδες που κυκλοφορούν ηλεκτρονικά, έτσι μέσω του διαδικτύου. Γιατί τότε η προσβασιμότητα των ε, μικρών ε, αυτών ε, εντύπων θα είναι προβληματική, δεν θα έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση, θα τους δυσκολευτεί στις πληροφορίες. Ξέρουμε ότι μερικές φορές πρέπει να πληρώνουμε για να έχουμε τέτοια πρόσβαση. Συνήθως δεν χρειάζεται να πληρώνουμε γιατί πληρώνει η διαφήμιση. Οι διαφημιστές όμως δεν θα πηγαίνουν τότε σε αυτούς τους μικρούς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάλτον εκ μέρου του ΙΣΙΑΡ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ όλους τους ομιλητές μας. Πρώτη ερώτηση. Γιατί βιαζόμαστε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί πρέπει τόσο γρήγορα να αποχωρήσουμε όταν δεν ξέρουμε ακόμα ποιε είναι οι επιπτώσει, ο αντίκτυπο του Γενικού Κανονισμού Προστασία Δεδομένων στι επιχειρήσει, που δεν έχουμε προλάβει να δούμε αν συμμορφώνονται. Δεύτερον, ποιο είναι το πρόβλημα, την Επιτροπή κύριε Ζώτα, ποιο πρόβλημα προσπαθούμε να λύσουμε. Εσεί Ευρωπαίοι τι λέτε, λέτε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό, το Skype, το έτσι και το άλλο, ναι, αλλά από την άλλη μεριά ανησυχούμε γιατί δεν προστατεύονται τα δεδομένα μα. Μα κοιτάξτε, Κανένα δεν έρχεται στην εκλογική μου περιφέρεια να μου πει θέλω να χρησιμοποιήσω το WhatsApp αλλά δεν μπορώ γιατί με προβληματίζει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πείτε μου για τα cookies. Τελικά πόσοι πηγαίνουν πίσω και λένε ναι στα cookies γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα. Έχει γίνει τέτοια ανάλυση. Και φτάνω και στο επόμενο έτσι. Το διαδίκτυο. Τι είναι. Έσοδα από τη διαφήμιση. Και ελεύθερη πρόσβαση. Δωρεάν. Τα cookies βοηθούν σε αυτό. Αλλιώς δεν θα υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες. Οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώνουν για κάτι που μέχρι τώρα ήταν δωρεάν. Οπότε αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποια έρευνα να δει πόσε τέτοιε δωρεάν υπηρεσίε θα χάσουν οι καταναλωτέ όταν περάσει ο κανονισμό αυτό. Και έχουμε και στην τέταρτη ερώτησή μου. Πώ θα ορίσετε τι συμπληρωματικέ υπηρεσίε για παράδειγμα για τα βιντεοπαιχνίδια που υπάρχει μια τέτοια έκθεση εδώ κοντά. Η ανακοίνωση αναφέρεται σε αυτά και θα συμπεριληφθούν τελικά στον κανονισμό και ποια θα είναι η επίπτωση του κανονισμού σε αυτά ή εξαρτάται από το ποιο θα είναι ο κανονισμός, ο ορισμός μάλλον που θα ισχύει για αυτές τις πληρωματικές υπηρεσίε, αν θα τα περιλαμβάνει ή όχι. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Χαλμπρέχτ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση. στην οποία θα ήθελα το δικό σας feedback. Αν δούμε το σημερινό νομικό πλαίσιο και την αναγκαιότητα που νομοθετούμε εδώ, δηλαδή το θέμα του απορρίτου επικοινωνιών και το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει της προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να πείτε ότι μπορούμε να έχουμε ένα λιγότερο προστατευτικό πρότυπο για τις τηλεπικοινωνίες και τα δεδομένα στο μελλοντικό κανονισμό από ό,τι έχουμε στη σημερινή νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Όταν απαντήσατε αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να μου πείτε πού βλέπετε η πρόταση ε, ουσιαστικά διατηρεί τα πρότυπα που βλεπετε η προταση ουσιαστικα διατηρει τα προτυπα που ειχαμε με τον προηγούμενο κανονισμό ή πρέπει να κάνουμε περαιτέρω δουλειά για να διατηρήσουμε το επίπεδο της προστασίας που έχουμε σήμερα υπό την οδηγία η privacy, κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της μέτρησης του ακροτηρίου στο διαδίκτυο και την συλλογή δεδομένων offline που μπορεί να γίνει κατά ε, την διάρκεια υπηρεσιών επικοινωνίας και συσκευών επικοινωνίας, της χρήσης συσκευών επικοινωνίας. Επίσης, θέλω να κάνω ένα σε ένα σχόλιο που ήδη έγινε όταν μιλάμε για τις ε, δωρεάν υπηρεσίες και το μοντέλο των δωρεάν υπηρεσιών σήμερα. Προφανώς ε, σήμερα κάποια επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται στην ε, αμοιβή που δίνεται μέσω της παρακολούθησης δεδομένων και της χρήσης των δεδομένων. Και αν αυτή είναι η πρόταση, θέτει αυτό σε κίνδυνο, αυτό μου υπενθυμίζει την ερώτηση πώς ακριβώς το σημερινό νομικό πλαίσιο αλληλεπιδρά με το επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στα δεδομένα και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες. Βλέπετε μια δυνατότητα σήμερα να έχουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο ε, βάση των δεδομένων που θα προέρχονται από τα δεδομένα των τηλεπικοινωνιών. Επειδή η κυρία Ζίπελ είναι η τελευταία μιλήτρια. Και δύο λεπτά. Παρακαλώ για να έχουν χρόνο και να απαντήσουν. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει δωρεάν υπηρεσία είτε πληρώνω με χρήματα, είτε πληρώνω με την ιδιωτικότητά μου. Και δεν θέλω σε κανένα να δίνω τη δυνατότητα να επισέρχεται στην ιδιωτική μου ζωή. Θα προτιμούσα να πληρώνω χρήματα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουταρέλη. Δεν είμαι σίγουρη αν ε, γνωρίζει ε, το πώς έχει φτιαχτεί η ιστοσελίδα της Γιώργο Άνοιξα αυτή την ιστοσελίδα στην αρχή της συνεδρίασης και κάτω-κάτω λέει ότι εργαζόμαστε με cookies. Συμφωνείτε? Και ε, Άλλο είναι όχι, αλλά δώσε μου περισσότερες πληροφορίες. Πάτησα λοιπόν το όχι, δώσε μου περισσότερες πληροφορίες. Και για μένα οι πληροφορίες που δόθηκαν δεν ήταν ιδιαίτερα επαρκείς. Έτσι λοιπόν άφησα τα πάντα, διέγραψα τις σελίδες από την εθονή μου και κάποιες, ε, κάποια λεπτά μετά ξανά άνοιξα τις σελίδες και τι έκπληξη ε, είχα τη σελίδα της Europol, αλλά όχι χωρίς αυτήν να χρησιμοποιούμε cookies. Έτσι λοιπόν η ερώτησή μου είναι, αυτή η ένδειξη, όχι δώσε μου περαιτέρω πληροφορίες, ερμηνεύτηκε ότι αφού διάβασα τις πληροφορίες συμφωνώ με τα cookies και τώρα έχω το cookie ή ερμηνεύεται όχι δεν συμφωνώ αλλά παρόλα αυτά μπορώ να δω την ιστοσελίδα. Μπορείτε να απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Uh, Μάλιστα, πολύ καλή ερώτηση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις εξαιρετικές ερωτήσεις συνάδελφοι. Τώρα να δώσω καταρχήν το λόγο στη Δέσποινα. Για 3-4 λεπτά παρακαλώ. Πολλές από τις ερωτήσεις πηγαίνουν προς την διακατεύθυνση, νομίζω. Και τον ε, ρώτησε, έρχεται καταναλωτές ε, που έρχονται και λένε δεν θα χρησιμοποιήσω την τάδε υπηρεσία λόγω των δεδομένων. Νομίζω ότι θα ακούσετε από τις παρουσιάσεις των καταναλωτών αργότερα ότι υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τη χρήση των δεδομένων. Δεν προσπαθούμε να σταματήσουμε την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να δώσουμε στους καταναλωτές ε, την δυνατότητα να μπορούν οι ίδιοι να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν και την κυριότητα των δεδομένων. Έχουμε μία πρόσφατη μελέτη η οποία έχει ένα τρομερό νούμερο, 92% αν θυμάμαι καλά, των πολιτών που ανησυχούν για το απόρριτο των δεδομένων τους. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλλά θέλουν και να έχουν την κυριότητα του τι συμβαίνει με τα δεδομένα τους, τον έλεγχο. Έτσι λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε, να τους ε, δώσουμε την προστασία που προβλέπει η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δηλαδή, όχι μόνο όταν λαμβάνουμε ένα γράμμα από την ταχυδρομία, αλλά όταν λαμβάνουμε και κάτι ηλεκτρονικά. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση της κυρίας Λάουρεστιν. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε στην πρότασή μας ήταν να δώσουμε μια επιλογή στους πολίτες. Να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων και η οδηγία υπέρβαση ε, προήλθαν ε, στα πλαίσια της ε, στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και υπάρχει εδώ μια κόκκινη γραμμή. Θέλουμε να δώσουμε καλύτερες επιλογές στους πολίτες, να μπορούν να ελέγξουν τι κάνουν και μπορούν να προσαρμοστούν σε εξελισσόμενα τεχνολογικά και επιχειρηματικά μοντέλα. Θέλουμε λοιπόν οι πολίτε να έχουν μια επιλογή και να μην ξεχνάμε ότι το λογισμικό δεν θα δουλέψει εκτό αν κάνουν μια επιλογή. Το σύστημα λοιπόν εξακολουθεί να προσφέρει απόρριτο εξ σχεδιασμού γιατί αν δεν επιλέξουν δεν μπορούν να πάνε παρακάτω. Και κάτι ακόμα, η πρόταση, ο κανονισμό δεν αποφασίζει για το αν θα πρέπει να το δεκτεί αυτό μια επιχειρήση ή όχι. Μπορείς να αποφασίσεις και ω επιχειρήση δεν θα προσφέρει την υπηρεσία σε κάποιον που θα κάνει μια άλλη επιλογή και δεν θα δώσει τα δεδομένα του. Είναι ελεύθερη αγορά. Αυτό είναι ο σχεδιασμός της πρότασης λοιπόν, έτσι όπως τη σκεφτήκαμε ως τώρα. Το ίδιο και για τη διαφήμιση. Η πρόταση δεν απαγορεύει τη διαφήμιση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρεξήγηση εδώ. Ούτε καθορίζουμε πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα επιχειρηματικά μοντέλα. Υπήρχε μια ερώτηση για την ανταλλαγή δεδομένων και για τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη συλλογή των δεδομένων. Υπάρχουν ήδη αυτά τα μοντέλα. Θα ξέρετε ότι έχουμε και μια άλλη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά δικαιώματα, σε ό,τι αφορά την περιοχή εγγύσεων. Θέλαμε να καλύψουμε και τα καταναλωτικά δικαιώματα όταν ε, τα ε, δεδομένα μας ζητούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή σε επιγραμμικό περιεχόμενο κτλ. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μας λοιπόν και εκεί το γεγονό ότι έχετε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε ανταλλαγή δεδομένων δεν σημαίνει ότι δεν έχει ε, δικαιώματα, είτε ω καταναλωτή, είτε δικαιώματα σεβασμού τη ιδιωτικότητα κτλ. Πολύ πρόσφατα ήμουν ε, σε ένα συνέδριο για τις ε, ε, κινητές ε, τηλεπικοινωνίες και βλέπω ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που αναπτύσσουν συστήματα που ανταμείβουν ε, τους καταναλωτές που αποφασίζουν να τους δώσουν τα δεδομένα τους και υπάρχει διαφάνεια για το ποια δεδομένα έχουν προσφέρει και τι παίρνουν ανταυτόν. Είναι ένας εξελισσόμενος τομέας λοιπόν. Και τι προσπαθούμε τώρα να κάνουμε για να απαντήσω σε άλλες πτυχές που ανέφερε και Θέλουμε ένα σύστημα που θα επιτρέψει στο να έχουμε ιδιωτικότητα και όχι να έχουμε σχεδιασμένα συστήματα. Ευχαριστώ, Τζοβάνι. Ευχαριστώ. Όταν ήμουν πρόεδρος πριν από 20 ε, χρόνια είχα ε, γράψει την ε, τελευταία εκδοχή της οδηγίας και ο στόχος είναι να μεταβούμε από τις αναλογικές στις ψηφιακές υπηρεσίες και αυτό αφορούσε τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών όμως. Με μερικούς μήνες αργότερα, ύστερα από την εφαρμογή, αρχίσαμε να αναλογιζόμαστε αν μπορεί να εφαρμοστεί και στο ίντρανετ αλλά και σε ορισμένε ε, υπηρεσίες διαδικτύου. Αν ε, μπορεί να εφαρμοστεί σε ε, δίκτυα και συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να ανανεώσουμε την οδηγία και στη συνέχεια μεταβήκαμε σε, μία, σε ένα νέο ορισμό αυτή τη φορά ή θέλαμε να υπάρχει συμφωνία με το συγκεκριμένο τομέα και αμέσως αρχίσαμε να έχουμε δυσκολίες αναλογιζόμενοι αν αυτό το νομικό πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί στο νέο φαινόμενο όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα, οι μηχανές αναζήτησης και πάλι για χρόνια είχαμε ερωτήματα ε, σχετικά ε, με, το, με την νομοθεσία και στη συνέχεια μεταβήκαμε στις ε, ε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τώρα επαφίεται στον κανονισμό να δούμε δούμε κατά πόσο ε, γίνεται σεβασμός των δικαιωμάτων μας. Ε, ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν οι κανόνες αυτοί ισχύουν, διότι υπάρχουν οι οποίοι γνωρίζουν τους κανονισμούς, αυτό το οποίο λέω είναι ότι ε, δεν είναι ξεκάθαρο και θα εκφράσουμε τις ανησυχίες μας αν όλες αυτές οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται ε, και θα πρέπει ίσως να επιλέξουμε διαφορετικούς ε, ή και πιο συγκεκριμένους κανονισμούς, κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε μεμονωμένα. Ε, διάβασα σε ένα tweet το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από 20 λεπτά ε, ότι υπάρχει ένα συμπέρασμα από έναν ειδικό ο οποίος ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση από τη ε, δική μου. Από τη δική μου. Και το δικό του συμπέρασμα λοιπόν ήταν εντελώς διαφορετικό. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη για να είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε ε, την 22 Μαΐου του 2018 διότι ε, η ε, υπάρχουσα οδηγία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η οποία δεν είναι σύμφωνη με το Γενικό Κοινωνισμό για την Προστασία Δεδομένων θα ε, πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα του, ε, του γνωμοδότη, ε, το οποίο είναι αναγκαίο όχι μόνο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά είναι ένα έτοιμα όλων των παραγόντων να αρχίσουμε ώστε να επιτρέψουμε στους ελεγκτές να μπορέσουν να εργαστούν με βάση αυτή την ημερομηνία. Τώρα όσον αφορά τους τομείς ανησυχίας, κύριε Άλμπρεχτ, ε, νομίζω ότι μπορούμε να ε, οικοδομήσουμε πάνω στους ε, τέσσερις βασικούς τομείς που αναφέρονται στην περίληψη και αυτό σχετίζεται ε, και ε, στην παρουσίαση του συναδέλφου μου, ε, το οποίο αφορά το Wi-Fi tracking για παράδειγμα, τους κανονισμούς με βάση τους οποίους το, η ανάλυση περιεχομένου και μεταδεδομένων θα επιτρέπεται και θα πρέπει να αναλογιστούμε την έγκριση όλων των τελικών χρηστών, αποστολέων και δεκτών και ε, τέλος ε, όσον αφορά ε, το tracking, η ομάδα εργασίας έβγαλε το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη αδειοδότηση από το χρήστη και τέλος αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να έχουμε την τις αυτόματες διατάξεις, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Τέλος, στο δικό σας ε, σχόλιο θα είμαι υπεύθυνος ε, ε, επέπτης από την 1η Μαΐου όσον αφορά τη Europol, θα ήθελα να σας διασφαλίσω ότι θα επιβάλλουμε, θα εφαρμόσουμε τους κανόνες όπως ορίζονται σε όλους τους θεσμούς της Ένωσης και αλλά και σε αυτόν τον ε, θεσμό εδώ στο κτίριο. Αν θέλετε να αναζητήσετε παραδείγματα, τότε θα μπορούσατε να μεταβείτε στην ανανεωμένη μας ιστοσελίδα ε, που ε, κυκλοφόρησε τέτοια στη λειτουργία την προηγούμενη εβδομάδα, όπου θα μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να εξαιρεθείτε, να έχετε ένα opt-out και θα σας δίνουμε όλες τις πληροφορίες, δεν παρακολουθούμε, τα ε, cookies είναι ε, σημαντικά για ορισμένες ε, υπηρεσίες και αυτό εξαρτάται από το πόσο βαθιά στην ιστοσελίδα μπαίνετε. Αν θέλετε να καταλάβετε όλη την νομοθεσία, τότε έχουμε, θα εκδώσουμε την οδηγία για αυτό που αφορά όλους τους θεσμούς και θα βασίζεται στα δεδομένα τα οποία έχουμε λάβει ως τώρα. όμως ε, πριν την 1η Μαΐου ε, θα ε, εμπιστευθώ τον επόπτη όπως και να έχει, είναι ένας τομέας όπου απαιτείται μεγαλύτερη διάβια και σεβασμός προς τους χρήστες από πλευράς όλων. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Ε, Δέσποινα, έχεις ε, να δώσει μια ακόμη απάντηση. Πολύ σύντομα, ο κύριος Άλπρεχτ είπε ε, πού μπορούμε να δούμε τις ε, διαφορές μεταξύ της υπάρχουσας οδηγίας και της, προ... και της πρότασης. Υπάρχουν τρία ξεκάθαρα σημεία. Πρώτον, δεν μιλάμε για μια οδηγία, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Μιλάμε λοιπόν για ένα κανονισμό. Δεύτερον, ε, η ε, βάση της συζήτηση είναι ότι ε, έχουμε τις επιφυείς υπηρεσίες, ότι τύπου δεν καλύπτονταν πριν και κάτι ακόμα το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά αναφερόμενη στον γενικό κανονισμό διότι στο υπάρχον σύστημα έχουμε ε, τέσσερις εκεί πάνω ε, υπηρεσίες που είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή με αποτέλεσμα να χάνουμε στην ορθή εφαρμογή λόγω ε, των δικαιοδοσιών που είναι πολύπλοκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να συμβεί Υπάρχουν προφανείς λοιπόν ε, λόγος, ε, λόγοι ε, για τα όσα κάνουμε και τις επιλογές που δίνονται. Και ο καθηγητής στο τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Θα επιλέξω μερικές. Αρχικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετές υπηρεσίες όχι δωρεάν αλλά online ε, χωρίς ακριβώς να πληρώνουμε με χρήματα. Ισχύει, όμως ε, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, ιδιαίτερως επειδή θα ακούσουμε αυτό το, επιχειρήμα, ε, αυτό το επιχείρημα αρκετά τον επόμενο, τον επόμενο χρόνο, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό χωρίς παρακολούθηση. Ε, για 100 χρόνια είχαμε το φωνό το οποίο ε, χρηματοδοτούνταν χωρίς να υπάρχει παρακολούθηση και θα ακούσουμε επιχειρήματα νέα όμως από τη δεκαετία του 90 και έπειτα έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα πληρωμής διαφημίσεων ε, το οποίο είναι αναγκαίο να παρακολουθούμε τους ανθρώπους online και επίσης θα ακούσουμε δεν λέω ότι το άτομο που έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα θα επιχειρηματολογήσει με αυτόν τον τρόπο όμως μπορεί και να ακούσουμε ότι ότι κάποιοι προτιμούν τις στοχευμένες διαφημίσεις διότι μπορεί να σχετίζονται περισσότερο με αυτό που θέλουν. Όμως αν κάτι τέτοιο ισχύει τότε δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, με την απαγόρευση των ε, τυχών παρακολούθησης διότι θα επιλέξει ο κόσμος τις στοχευμένες διαφημίσεις. Όμως δεν υπάρχουν απαγορεύσεις, ε, υπάρχει στην πρόταση το ζήτημα της της έγκρισης. Ε, επίσης όλο αυτό δεν λέει τίποτα για τις ε, διαφημίσεις. Κυρία Αλμπρέχτ, ε, ρωτήσατε για την μέτρηση των χρηστών. Όσοι δεν γνωρίζουν καλά την πρόταση, αναφέρεστε στην ανάγκη ε, έγκριση των cookies με κάποιες εξαιρέσεις όπως είναι τα cooking για το login ή για ε, ε, τις αγορές. Είναι κατά βάση μια καλή ιδέα, όμως υπάρχει μια εξαίρεση σχετικά με την μέτρηση των χρηστών. Σύμφωνο ότι για ορισμένα cookies ιδιωτικότητα θα πρέπει να υπάρχει ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη έγκρισης, όμως ε, για κάποια cookies που είναι ουδέτερα εκεί θα πρέπει να ορίζεται ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Υποστηρίζω μία εξέρεξη, μία εξέρεξη στα συγκεκριμένα cookies, όμως αυτό θα πρέπει να οριστεί καλύτερα. και θέσατε ένα ακόμα ερώτημα σχετικά με τη συλλογή των offline δεδομένων όπως είναι ε, για, περί, για παράδειγμα ε, τις ε, κονσόλες παιχνιδιών οι οποίες ε, καταγράφουν οι ε, τηλεοράσεις οι οποίες μπορεί να ενεργοποιούνται και να παρακολουθούν. Βέβαια υπάρχουν υπηρεσίες όπως είναι οι αγορές online. Όντως όλο αυτό δεν ορίζεται στην πρόταση, θα πρέπει να το αναλογιστώ. Όμως ναι, ο κανονισμός θα πρέπει να ε, ε, προστατεύει την ιδιωτική ζωή την οποία τη βιώνουμε στο σπίτι μας και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχει νόημα να εισαχθούν ε, κανόνες σχετικά με το ίντερνετ των πραγμάτων που μπορεί να αρχίσουν να παρακολουθούν ξαφνικά μέσα στο σπίτι σας. Και τέλος όσον αφορά το ερώτημα της κυρίας Λαριστίν ε, βλέπετε τους ε, μαύρους κύκλους ε, στα μάτια μου, οπότε δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό το πλάνελ. Θα μπορούσαμε να ρωτάμε ξανά και ξανά, αλλά δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Φεντερίκ, Τζοβάνι, Δέσποινα. Σας ευχαριστώ για τις παρουσίες σας και τις απαντήσεις σας. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Περάστε παρακαλώ εδώ. Στο μεταξύ εγώ θα κάνω την εισαγωγή. Θα μιλήσουμε για την νομική συνέπεια της πρότασης αυτής με τα υπόλοιπα ε, νομικά μέσα και εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Δύο είναι, κυρία, οι στόχοι της πρόταση της Επιτροπής, η συνέπεια, όπως σας είπα, αλλά και η επίσης όρης εφαρμογή των ε, προτινόμενων μέτρων. Η συγκίτρια βλέπω βγαίνει, αλλά φαντάζομαι θα επανέλθει. Θα ακούσουμε εκπροσώπους της, ε, των τηλεπικοινωνιών, του διαφημιστικού κλάδου, από τον ακαδημαϊκό χώρο. Έχουμε τέσσερις ομιλητές. Καθίστε παρακαλώ όλοι εδώ και τρίστε το χρόνο σας για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε, ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο Αντώνιο Μάρκος, ο οποίος είναι σύμβουλος καταναλωτών στην τηλεφώνικα για τα μεγάλα δεδομένα. Θα μας δώσει λοιπόν την οπτική γωνία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Παρακαλώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Οι φορείς των τηλεπικοινωνιών πάντα ενδιαφέρονταν για την ασφάλεια και την προστασία του ιδιωτικού βίου των τηλεπικοινωνιών στα διάφορα δίκτυα. Και αυτό αποτελεί και το κύριο στοιχείο που μας καθοδηγεί στις επιλογές μας όταν δραστηριοποιούμεθα. Για παράδειγμα, συμμετέχουμε στις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα μεγάλα δεδομένα είναι ένα παράδειγμα προσπάθειας που γίνεται από και διαφορετικές χώρες, συγχρόνως με ακαδημαϊκούς και με τον κλάδο, για να σεβόμαστε τον ιδιωτικό βίο και να προστατεύουμε τα δεδομένα στο, στην περιαγωγή. Πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία για όλες τις ε, πλευρές. Τις τηλεπικοινωνίες, τους παρόχους πληροφοριών, τους καταναλωτές και τις εποπτικές αρχές. Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Δεδομένων προτάθηκε για την προστασία του ιδιωτικού βίου και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται. Προτείνει εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές διαδικασίες, διαφορετική χρήση και διαφορετικές επιθυμίες προστασίας. λογοθεσία, οι επιπτώσεις, η προστασία του ιδιωτικού βίου βάσει σχεδιασμού, συμβατότητα, πολλές δυνατότητες, επιλογές. Όλα αυτά πρέπει να συνάδουν με την προστασία του ιδιωτικού βίου και την νομική προστασία. Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την εκπόνηση κανόνων προστασίας όσον αφορά τα μεταδεδομένα και τις τηλεπικοινωνίες. Κανόνες που να είναι συνεπείς με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και καινοτόμες μεθόδους στη χρήση δεδομένων. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι σε έναν κόσμο επικοινωνίας όπως είναι ο δικός μας, τα περισσότερα δεδομένα ε, συνδέονται με τις επικοινωνίες. Τώρα για το θέμα της ε, ισότιμης μεταχείρισης. διαφορετική μεταχείριση δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιπτώσεις που δεν συνάδουν με αυτά τα οποία θέλουμε. Τα μέτρα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα πλαίσια, σε εντοπισμό και τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν με τα δεδομένα και τα δίκτυα θα μπορέσουν έτσι να τα εκλάβουν σαν δεδομένα προς χρήση από τα δίκτυα παρόχων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είχε κακές συνέπειες αν φτάνανε σε λάθος χέρια. γιατί τα ίδια δεδομένα μπορεί να τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα με το ποιοι συμμετέχουν στην αλυσίδα αξιολόγηση. Το θέμα τώρα της συνένεσης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι αδιαφεσβήτητο ότι πρέπει να υπάρχει. Αλλά διαφορετικές ε, αιτίες που μας οδηγούν στην προστασία πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εκπονούμε τους κανόνες για την προστασία των ε, δεδομένων. Αυτό το λέει και η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναζητούμε την προστασία δεδομένων γιατί εξαρτάται από το τι αντίκτυπο θα έχει στις τηλεπικοινωνίες τους. Συνεπώς, η αρχή λογοδοσία του Γενικού Κανονισμού Προστασία Δεδομένων πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε φορά που μιλάει και για μέτρα άμβληση. Να υπάρχουν ε, αντιμηχανισμοί, εξαιρεσει κυρίως τεχνικές οι οποίες να εξηγούν πόσο μεγάλη σημασία έχει η προστασία των δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Συγχρόνως, να προστατεύεται ο ιδιωτικό βία. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα μεγάλα δεδομένα αναγνωρίζει τα στοιχεία αυτά. Η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και η κυκλοφορία τους είναι κάτι από το οποίο μπορούν να υποφεληθούν για παράδειγμα αρχές μεταφορών. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την κοινωνική ή ακόμα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, στις μεταφορές, στην εκπαίδευση, στην υγεία, ε, στις οικονομικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο κλπ. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Εδώ τα δίκτυα έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η επεξεργασία των μεταδεδομένων είναι σημαντική όχι μόνο για την ασφάλεια των δικτύων, αλλά και για την ασφάλεια των φορέων, των συστημάτων και των υπηρεσιών των παρόχων. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την οδηγία ΕΝΕΣ και γι' αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε την συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια των δικτύων. Η συνεργασία αυτή πρέπει να γίνει και στον τομέα της επεξεργασίας ε, των δεδομένων. Το ίδιο και για τις απάτες που μπορεί να γίνονται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αλλά και στην συμπεριφορά που επηρεάζει τρίτα μέρη. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασία Δεδομένων λαμβάνει υπόψη και αυτή τη διαδικασία. Επίσης, στατιστικά δεδομένα, ανάλυση μεταδεδομένων όταν δεν επηρεάζεται ο ιδιωτικό ο βίος πρέπει να εξεταστεί για το κατά πόσο είναι κάτι που συνάδει με, τη, με ό,τι έχουμε μέχρι τώρα ή όχι. Οι εξαιρεσει δεν θα βοηθήσουν απαραίτητα να υπάρχει η κατάλληλη ευελιξία. Υπάρχει το άρθρο 6, σημείο 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασία Δεδομένων που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για όλα αυτά. Ο τρόπος που γίνεται επεξεργασία, οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, οι προσδοκίες των καταναλωτών, όλα αυτά οδηγούν σε μια νοοτροπία προστασίας των δεδομένων. Και από εκεί πρέπει να απορρέει και η τελική ρύθμιση Τέλος, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητε επεξεργασίας μεταδεδομένων που δεν επηρεάζουν την, τον ιδιωτικό βίο ή την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Γκριμτάλ, ο οποίος ε, θα μας ε, δώσει την ε, σκοπιά από τον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα το απόγευμα και θα ξεκινήσω με δύο λόγια ε, για τη ΣΥΠΣΤΕΤ. Είμαστε μία από τις ηγετικέ επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη. Έχουμε δραστηριοποίηση σε επιγραμμικές επιχειρήσεις, ε, στα μίντια, σε επιγραμμικές σημεία πώληση και έχουμε θέσεις στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και τη Σουηδία. Ουσιαστικά ένα ακριβώς λίθος του επιχειρησιού μα είναι ε, τα μέσα για τι ειδήσει. Έχουμε διάφορε ιστοσελίδε για τι ειδήσει ε, και την Aftonbladet ε, που είναι η κύρια ιστοσελίδα. Ο προτινόμενος κανονισμός είναι πολύ σημαντικός. Θα πλήξει αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας, την ικανότητα των ευρωπαϊκών εταιριών να ανταγωνιστούν με τους παγκοσμίους παίκτες και τέλος πρόκειται για τη δημοκρατία η πρόταση μπορεί στην πραγματικότητα να έχει επίπτωση ε, στον ε, ανεξάρτητο και δωρεάν ευρωπαϊκό τύπο σε μεγάλο βαθμό. Μόλις πριν λίγα χρόνια οι κύριοι ανταγωνιστές μας ήταν άλλες ε, τοπικές εταιρείες. Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε τεράστιο και ξενόμενο ανταγωνισμό από τους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες. Τώρα είναι ζωτικό να υπάρξουν κανόνες που θα διασφαλίσουν ίσους κανόνες για όλους. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα ο κλάδος μας ξέρει πολλά μοντέλα επιχειρηματικά. Ε, έχουμε, παραδείγματο χάρη, πρόσβαση στο περιεχόμενο επιπληρωμή και δωρεάν περιεχόμενο με διαφήμιση. Ε, βλέπουμε από μία μελέτη που κάναμε ότι δέχονται οι καταναλωτές μας σε μεγάλο βαθμό τις διαφημίσεις όταν ε, δεν ενοχλούν. Ε, μόνο το 20% ε, των εσόδων των εκδοτικών οίκων έρχεται από την πληρωμή των χρηστών. Αυτό μας δείχνει ότι η ύπαρξη του ελεύθερου, του δωρεάν τύπου στην Ευρώπη που είναι προσβάσιμο στο κοινό εξαρτάται από την ικανότητά μας να έχουμε ε, δωρεάν διαφήμιση. Μάλλον, συγγνώμη, να δούμε αποτελεσματική διαφήμιση. Σήμερα περίπου το 60% της ψηφιακής διαφήμισης στη Σουηδία πηγαίνει στο Facebook και στο Google και συνεχώς αυξάνεται το μεριδιό του στην αγορά. Σε άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Συνδέεται η ισχυρή του θέση με την πρόσβαση στα δεδομένα, ε, τα οποία δεδομένα είναι πολύ πιο πολύτιμα ε, αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου είναι ότι οι παγκόσμιοι παίκτες είναι σε καλύτερη θέση για να σεβαστούν τους προτινόμενους κανόνες. Οι εκδότες, σε αντίθεση με τους παγκόσμιους παίκτες, εξαρτώνται από τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την ε, παρουσίαση διαφημίσεων. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι ε, μεγάλες εταιρείες όπως η Groom ε, M, Red Media κτλ. Ε, διάφοροι πολιτές τεχνολογίας όπως η AppNexus ε, ή διάφορες πλατφόρμες για να αναφέρω ορισμένε. Οι παγκόσμιοι παίκτες μπορούν να κάνουν τα πάντα in-house, εντός και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τρίτα μέρη για να τους βοηθήσουν σε αυτές τις διαδικασίες. Η πρόταση περιορίζει την χρήση πολιτών τρίτων μερών και εταίρων. Δηλαδή, τι θα γίνει στην πράξη είναι ότι η πρόταση αυτή ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τους μεγάλους παγκοσμίους παίκτες. Προκειμένου να ανταγωνιστούμε με τους ε, παγκόσμιους παίκτες, ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ανεξάρτητο ευρωπαϊκό τύπο και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ψεύτικες ειδήσει, χρειαζόμαστε δεδομένα και γνώση για όσους χρησιμοποιούν τις επιχειρήσεις μας. Πρέπει να μάθουμε για τη συμπεριφορά τους και τα ενδιαφέροντά τους ε, τι θέλουν. Μόνο με αυτή τη γνώση μπορούμε να παράσχουμε πρόσωποποιημένο περιεχόμενο και προϊόντα. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις είναι όσο δυνατόν ε, πιο στοχευμένες, ότι εμφανίζονται ε, στα, ε, τη σωστό χρόνο στους ανάλογους καταναλωτές και τα λοιπά, χρήστες και τα Φυσικά τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά στο πλαίσιο της διαφήμισης, όμως τα δεδομένα είναι ζωτικά και για την ανάπτυξη του προϊόντος μας και προκειμένου να παράσχουμε προσωποποιημένες εμπειρίες online. Μπορώ να αναφέρω ότι στη ΣΥΠΣΤΕΤ τώρα οικοδομούμε μια νέα πλατφόρμα όπου η προσωπικοποίηση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά. Αν οι καταναλωτέ μα δεν μα εμπιστεύονται, τότε δεν θα μα επιτρέψουν ε, να έχουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του. Επομένω, είναι απλό για μα. Χρειαζόμαστε δεδομένα Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές μας μας εμπιστεύονται. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην καινοτομία ε, του ιδιωτικότητα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, να κοινοποιήσουμε με σαφήνεια πώς και γιατί συλλαγούμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας. Δεν θα είναι δυνατό οι χρήστες ε, να κατανοήσουν πότε ουσιαστικά κατεβάζουν πράγματα από έναν φιλομετρητή. Και είναι πολύπλοκα όλα αυτά. Δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι οι καταναλωτέ κατανοούν τα πάντα και παίρνουν ενεργή στάση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές αποτελεσματικά μπορούν να κάνουν επιλογές ε, για το πώ χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του. Εμείς ε, ουσιαστικά χτίζουμε ένα εργαλείο ιδιωτικότητα για να το διευκολύνουμε αυτό. Βλέπετε τώρα στα αριστερά σα ε, ε, κάτι τέτοιο. Πρόκειται για μια επένδυση για να διασφαλίσουμε ότι κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για του καταναλωτέ. Επομένω, για να συνοψίσω. Νομίζω ότι το opt-in δεν είναι η λύση. Είναι ένας πολύπλοκος ε, τομέας αυτός δεν μπορούμε να έχουμε την ε, βασική προσδοκία ότι οι καταναλωτές κατανοούν και τοποθετούνται ενεργά και διαλέγουν το opt-in. Ε, επίσης, ούτε νομίζω ότι το opt-in πρέπει να γίνεται μέσω των φιλομετρητών, ε, γιατί διαφορετικά με αυτόν τον τρόπο θα είναι οι φιλομετρητές οι φύλακες του διαδικτύου και αυτό δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των καταναλωτών και μην ξεχνάτε ότι πολλοί από τους φιλομετρητές είναι ανταγωνιστές μας. Παίρνουν το σχάρι, το Google Chrome, ε, το Safari της Apple, όλοι αυτοί είναι φιλομετρητές. Επίσης δεν είναι η κατάλληλη απάντηση να προσπαθήσουμε ε, να βάλουμε το θέμα της διαφάνειας και της ενδυνάμωσης του χρήστη ε, με μία και μόνη λύση. Πρέπει να έχουμε αντίθετα ευέλικτους κανόνες που να διασφαλίζουν ίσους κανόνες ανταγωνισμού και να επιτρέπουν την καινοτομία σε ό,τι αφορά στο θέμα του σεβασμού του απορρίτου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φάνη Χετβέγγι είναι η επόμενη ομιλήτρια και εκπροσωπεί μία ΜΚΟ, την Access Now, η οποία ουσιαστικά υπερασπίζει τα ψηφιακά δικαιώματα των χρηστών σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Ονομάζομαι Φανή ε, Χίτβεγκη. Ε, προέρχομαι από μία ΜΚΟ με έδρα της Βρυξέλλες, ονοματιάξης ΝΑΟ και όπως έχει πει ο Πρόεδρος, Στόχος μας ε, είναι ε, να ε, υπερασπιστούμε τα ψηφιακή δικαιώματα των Χριστών σε όλο τον πλανήτη και θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα για, την, για τον προτινόμενο κανονισμό. Ο τίτλος αφορά την νομική συνέπεια της, ε, του συγκεκριμένου ε, κανονισμού. Στόχος μας είναι να ε, τηρήσουμε τους κανονισμούς της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και να ακολουθήσουμε τη νομική συνοχή με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Η Access Now καλωσορίζει λοιπόν την προσπάθεια της Κομισιόν να μεταρρυθμίσει τους κανονισμούς της e-Privacy και να συγκεκριμενοποιήσει τον Γενικό Κανονισμό. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος κανόνες ε, δεν θα πρέπει μονάχα να τηρούν το επίπεδο προστασίας το οποίο ορίζεται από το γενικό κανονισμό αλλά ταυτόχρονα να το ξεπεράσουν για να προστατεύσουν ε, το ε, δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Όπως ορίζεται από το άρθρο 29 της ομάδας εργασίας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα όλο αυτό δεν ακολουθεί τις συγκεκριμένες υποσχέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα επιχειρήματα των διαφόρων παραγόντων ε, συνήθως έχουμε τις δύο αντικρουόμενες απόψεις οι οποίες αφορούν το ίδιο το οποίο είναι είτε να γίνουν πιο αυστηροί οι κανονισμοί ή πιο χαλεροί. Άλλοι λένε ότι ε, ο γενικός κανονισμός είναι μια χαρά ε, όσο έχει παρά τις, προ... τις πρώτερες προσπάθειες ε, να δημιουργηθούν προβλήματα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι ο γενικός κανονισμός ήδη δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Προσωπικά διαφωνώ και με τα δύο επιχειρήματα και παρόλο που χαιρετίζω το, την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γενικό κανονισμό, θα ήθελα να πω ότι δεν διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και το απόρριτο τη επικοινωνία και δεν προσφέρει αρκετέ προστασίε όσον αφορά το, την, ε, το online, ε, την online παρακολούθηση και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αυτή τη μεταρρύθμιση. Δεύτερον, να αρνούμε το χαρακτηρισμό ότι είναι υποχρεωτικό ο γενικό κανονισμό για να σεβαστούμε τα συγκεκριμένα ε, δεδομένα, τα, τα συγκεκριμένα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε. είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να ορίζεται από τους χρήστες και για να υπάρχει η νομική συνοχή με το γενικό κανονισμό θα πρέπει να στοχεύσουμε στα κάτωθη. Ε, αφενός, ε, ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να έχει δεσμευτικό και απαιτήσει ε, τόσο για τους παρόχους hardware και software. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη ε, προστασία για το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το εύρος των μεταδεδομένων και να αναγνωρίσουμε ε, τις ευαίσθητες πληροφορίες. Επίσης το εύρος βασίζεται σε δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αφορά τόσο τα μεταφερόμενα δεδομένα αλλά και αυτά τα οποία αποθηκεύονται. Επίσης, ε, η έγκριση ε, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και βάσει τη ευαισθησία των δεδομένων τα οποία προστατεύονται από τον κανονισμό ε, του e-privacy δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, ως ευκαιρία για την επεξεργασία. Και τέλος θα πρέπει να ορίζονται, να ορίζονται ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τους συγκεκριμένους κανονισμούς και θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση και από τις ΜΚΟ η συμφωνία με το γενικό κανονισμό θα οδηγήσει σε μια ισότιμη συμμετοχή. Ε, βέβαια αυτή η έννοια χρησιμοποιείται ε, παρασάγκας με αποτέλεσμα να ξεφεύγουμε δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε ε, για το OTT μονάχα, για τις επιφύγεις υπηρεσίες. Ε, το, ε, η ισότιμη συμμετοχή θα πρέπει να υπάρχει για την προστασία των καταναλωτών, διότι είναι άνηση. Οι ε, πάροχοι λοιπόν έχουν ε, μια ηγετική θέση όσον αφορά τη διαφάνεια ε, και τη συνοχή και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασυνέπεια. Θα πρέπει λοιπόν ο κανονισμός να επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας ασχέτως των υποδομών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα αλλά όχι για τους ορισμούς που χρησιμοποιούν οι Βρυξέλλες για τις διάφορες εφαρμογές και συσκευές όπως ε, λέει η ημερήσια διάταξη της ακρόασης, ε, θα πρέπει ε, να επικεντρωθούμε στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να διασφαλίσουμε το ίδιο επίπεδο προστασίας για άτομα ασχέτως των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται και φοβάμαι ότι αυτό δεν γίνεται. Ο ορισμός των κανονισμών δεν θα πρέπει να επαφίεται στον στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ε, διότι ε, κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα, διότι δεν επηρεάζει τη μεταρρύθμιση ε, του e-privacy και δεύτερον δεν είναι ξεκάθαρος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το περιεχόμενο επίσης θα πρέπει να είναι πιο περιεκτικό και ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει βάση για την συγκεκριμένη πρόταση Έχουμε ένα πρόσφατο ε, παράδειγμα σχετικά με το πώς ε, έγινε άφηση των συγκεκριμένων κανονισμών. Έχουμε το 92% των ανθρώπων ε, οι οποίοι επιθυμούν να υπάρχει το απόρριτο των επικοινωνιών τους σύμφωνα με το βαρόμετρο του 2016 και αυτή είναι η ευκαιρία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραδώσει. Όμως η πρόταση ως εκ τούτου θα πρέπει να αυξήσει ε, το επίπεδο προστασίας ε, για να ε, παρέχει καλύτερη προστασία από ότι ο γενικός κανονισμός, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ισότιμη συμμετοχή για όλους τους παράγοντες, ιδιωτέρως για τους χρήστες, οι οποίοι, στους οποίους έχουμε υποσχεθεί ότι θα δοθεί ο έλεγχος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, η οποία θα είναι επιτυχημένη μονάχα σε περίπτωση που ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο τελευταίος ομιλητής μας είναι ο καθηγητής Ράνενμπεκ, ο οποίος ε, είναι ο ε, επικεφαλής ε, της έδρας online ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο Γκέτε της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζουμε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας στην ακρόαση αυτή. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τις διάφορες οργανώσεις, του διάφορους συμβούλους. Δεν είναι ο κατάλογος βέβαια πλήρης, αλλά όλοι αυτοί συνεισφέρουν στον προβληματισμό μας και θέλω να τους ευχαριστήσω. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ θέλω να αναφερθώ λίγο στο παράδοξο ότι των προστατευμένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ανάγκη της προστασίας και με την αγορά των OTT, των over the top, των επιπλέον των πρόσθετων υπηρεσιών και την ανάγκη να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες. Πρέπει να δούμε πού βρίσκονται τα δεδομένα, ...πώς γίνεται η ανείχνευση Bluetooth κλπ. Επόμενη διαφάνεια. Τι εννοώ με αυτό το παράδοξο, την προστασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. επικοινωνίε. Οι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε χρειάζεται να προστατεύονται όλο και περισσότερο για να προστατεύεται το απόρριτο ιδιωτικό βίο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από την αγορά. Οι τηλεπικοινωνίε που δεν είναι προστατευμένε είναι δωρεάν ο κανονισμό μέχρι τώρα καλύπτει ένα τμήμα τη αγοράς μόνο, τι παραδοσιακές και δεν υπάρχει και ισότιμη αντιμετώπιση. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι και να συμπεριληφθούν αυτές οι over the top τηλεπικοινωνίες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να γίνει. Η προστασία των λεπικοινωνιών είναι σημαντική και όπως είπαν και οι προηγούμενοι δεν πρόκειται μόνο για ένα προσωπικό δικαίωμα ιδιωτικό αλλά πρόκειται και για την ίδια την λειτουργία της δημοκρατίας και άρα πρέπει να πάμε λίγο πιο μακριά από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Τι γίνεται στην αγορά τώρα. Οι υπηρεσίε τηλεπικοινωνιών ήταν μέχρι τώρα από μόνο του ένα καλό προϊόν που πουλιόταν, είχε την τιμή του. Σήμερα όμως οι ότι προσφέρουν δωρεάν τηλεπικοινωνίες και ανταγωνίζονται τους ε, παράγοντες στην αγορά που είχαμε μέχρι τώρα. Εδώ αναφέρονται κάποια παραδείγματα. Οι τιμές επίσης μειώνονται και μειώνεται και η ποιότητα, μειώνεται και η εμπιστοσύνη και τελικά οι καταναλωτές δεν έχουν εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους προϊόντα και το να μην προστατεύονται οι τηλεπικοινωνίες είναι πολύ κακό και για την ίδια τη δημοκρατία. Ο κανονισμός λοιπόν λέει ανεξάρτητα από την πληρωμή και θέλει όλο και περισσότεροι παίκτες να καλύπτονται. Αυτά όλα όμως δεν φτάνουν και γι' αυτό θέλω εδώ να σας παρουσιάσω λίγο τις αγορές OTT. Εδώ ίσως δεν υπάρχουν όλα, πάντως το βασικό είναι ότι μια παραδοσιακή αγορά OTT έχει επενδυτές που θέλουν να έχουν όσο γίνεται περισσότερους χρήστες, να υπάρχουν, ε, τα ξέρει ποια είναι τα προφίλ, να χρησιμοποιούνται και εδώ δεν πρόκειται μόνο για τους καταναλωτές, είναι κάτι που πουλιέται ευρύτερα. Συγχρόνως όμως η εφαρμογή δεν καθορίζεται απόλυτα. Υπάρχει το Facebook, υπάρχει το Google. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να υπάρχει μια τάση κυριαρχίας της αγοράς από λίγους μόνο παίκτες οι οποίοι διαθέτουν την πηγή των δεδομένων. Μπορούν έτσι να προστατευτούν οι συνταγματικές αξίες. Χρειάζονται καλύτερα προστατευμένες υπηρεσίες, άρα με παίκτε οι οποίοι να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη προστασία. Τι εννοούμε συγκεκριμένα για τα OTTs. Να λοιπόν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δεδομένο της τοποθεσίας, το που βρίσκεται κανείς, ο εντοπισμός του και τι στοιχεία μπορεί κανείς να έχει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν, βλέπετε, είναι τα διάφορα σενάρια που έχουμε στα offline, online. Έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, δεν τα βλέπουμε βέβαια όλα. Πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε στο μετανορισμό των μεταδεδομένων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, τα άρθρο 4, τα άρθρο 8. Το 4 έχει τον ορισμό των μεταδεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν προσφέρουν ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες. Αυτό όμως σαν ορισμός είναι πάρα πολύ στενός γιατί δεν καλύπτει τις υπηρεσίες over the top. Άρα υπάρχει περιορισμένη προστασία για τους καταναλωτές. Είναι δύσκολο οι καταναλωτές να εμπιστευτούν λοιπόν τέτοια δεδομένα και είναι ένα μειονέκτημα και για τους ίδιους τους παρόχους. Αυτό πρέπει να αλλάξει και η πρότασή μου είναι να υπάρξει ευρύτερη προστασία και περισσότερες, περισσότερες ότιμες συνθήκε. Εδώ έχετε έναν χάρτη θερμότητας. Πρόκειται για ένα geospatial clustering. Κάποιοι είναι στην Βαρκελόνη το σημείο 17 λέει ότι πρέπει να βρεθούν αυτοί οι οποίοι εντοπίζουν, τα, οι μηχανισμοί οι οποίοι εντοπίζουν. Η μετακίνηση για να μπορούμε να αποφεύγουμε μποτιλιαρίσματα. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον να εντοπίζονται. Και κυρίως αν υπάρχει μια ολόκληρη σειρά μεταδεδομένων. Μπορεί δηλαδή να εντοπίσει ο μηχανισμός που βρίσκεται ένας τουρίστας και που βρίσκεται μετά από 5 λεπτά. Μπορεί να γίνει αυτό ακόμα και χωρίς ψευδόνυμα. Πρέπει να αλλάξει η αναφορική σκέψη 17. Τώρα το άρθρο 8β, στο 2β στο οποίο αναφέρθηκα πριν, συλλογή ζωνών με εντοπισμό Wi-Fi και Bluetooth οι καταναλωτές, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε μια ζώνη όπου μπορεί να εντοπιστεί το Wi-Fi, το Bluetooth. Δεν έχει να κάνει αυτό δηλαδή με τη τηλεφωνία, έχει να κάνει καθαρά με υπηρεσίες over the top. Και πρέπει να κλείσει κανείς το κινητό του αφού δει ένα μήνυμα που βγαίνει, μια προειδοποίηση. Αλλά ο εντοπισμό αυτός μπορεί να γίνει χωρίς συνένεση από τον ενδιαφερόμενο. Εμείς θέλουμε προωθημένες υπηρεσίες, τι κάνουμε, μπαίνουμε και κοιτάμε και ψάχνουμε, υπάρχει κάπου προειδοποίηση όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο για να ξέρω αν πρέπει να κλείσω το κινητό μου ή όχι. Δεν νομίζω ότι κανείς συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν αυτά είναι πράγματα τα οποία λείπουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων δεν υπάρχει σύνδεση στο άρθρο 21 με το άρθρο 80 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε είναι να μην είναι πάντα υπεύθυνο ο πελάτης. Το άρθρο 8 και 10 πάνε πέρα από τις ταμπλέτες και τα κινητά. Έχουν να κάνουν με παντός είδους software το Internet of Things που μπορεί να είναι ας πούμε το, το μου Πρέπει να δω με τι συνδέεται και κατά πόσο μπορεί κανείς να ξέρει τι μηχανήματα έχω εγώ, τι φωτοτυπικά μηχανήματα. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα. Να, πώς μπορεί κανείς να έχει δεδομένα. Από την ε, καφετιέρα μου, για παράδειγμα, ή από το ξυπνητήρι μου. Όλα αυτά συνδέονται με το διαδίκτυο. Και να και κάποια άλλα με το Bluetooth που συνδέονται. Να και άλλα. Ζυγαριά και λοιπά. Όλα αυτά μπορούν ε, να είναι μηχανήματα στα οποία έχουμε πρόσβαση από το διαδίκτυο. Να και κάποια άλλα. Γι' αυτό όλα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό. Και άλλα, και άλλα, επόμενο, Το σπίτι μας, να κάποια άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Και το τελευταίο που μόνο στην Ιαπωνία υπάρχει, τουαλέτα, το καζανάκι. Μπορεί να συνδεθεί και αυτό με το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Toilets are in Europe. Μάλιστα, ευχαριστώ. Εμεί ε, ε, έχουμε και άλλε τολέτε στην Ευρώπη που έχουν διαφορετικά καζανάκια. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ όλους για το χρόνο σας. Ακούσαμε ουσιαστικά τις ΜΚΟ, τον κλάδο της διαφήμισης, τον εθνική τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Έχουμε λίγο καθυστερήσει όμως με το χρόνο. Προσπαθήστε παρακαλώ να είστε σύντομοι συνάδελφοι και να ξεκινήσουμε και πάλι με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ήταν ε, πάρα πολύ πλούσιες οι παρουσιάσεις και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει ε, και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαζόμασταν, μάλλον τέσσερι ώρε για να κάνουμε μια πλήρη συζήτηση. Τέλο πάντων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μαζικά δεδομένα. Αναφερθήκατε σε μια έκθεση, όμως στην έκθεση θα πρέπει να εφαρμόζεται η προστασία των δεδομένων ε, και σε αυτόν τον ε, τομέα. Αυτό ήταν κάτι γενικό. Τώρα, αν δούμε τον κανονισμό, η privacy και τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμη κάποια μαύρα σημεία. Εγώ να σας πω ποια είναι η δική μου εντύπωση, να μου πείτε ίσως αν έχω δίκιο ή άδικο αισθάνομαι ότι επικεντρωνόμαστε περισσότερο στη συλλογή προσωπικών δεδομένων σαν συνεισφορά για την ανάλυση δεδομένων και λιγότερο μιλάμε για τη χρήση ή για τα αποτελέσματα. Όμως ε, αυτά τα δεδομένα μπορεί να μην είναι προσωποποιημένα, μπορούν, ε, παίρνουν το σχάρι, να ληφθούν από αλλού. Δεν είναι όμως πολύ σαφή τα πράγματα, δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες, ε, ούτε στην e-privacy σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των δεδομένων που μέσω της αναλυτικής ε, γίνονται προσωπικά δεδομένα ενώ όταν συλλέχθηκαν στην αρχή δεν ήταν προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, ε, αυτό δεν έχει να κάνει με την επεξεργασία στη στάδια πριν από τη χρήση. Ίσως ε, να χρειαζόμαστε και διαφορετική διατύπωση εδώ Μήπως ε, θα μπορούσατε να μας πείτε ποια διατύπωση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντικατοπτρίσουμε την ιδιαιτερότητα της αναλυτικής των μαζικών δεδομένων. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση. Να σχολιάσω. Στις επαφές με την ενδιαφερόμενα μέρη δεχτήκαμε πολύ πίεση από τον τομέα των εκδόσεων. Είχαμε κάποιες ε, ε, κάποιες θέσεις ε, ουσιαστικά που μας μιλούσαν σαν έρχεται το τέλος του κόσμου, ότι σκοτώνουμε τώρα τον κλάδο των εκδόσεων. Πού βλέπετε να είναι αυτές οι κοκκινές γραμμές. Τι είναι τόσο σημαντικό που χωρίς αυτό δεν ε, μπορείτε να τυπώσετε τίποτα. Γιατί εμείς ε, είδαμε βάσει των ε, ερευνών μας ότι μπορείτε να έχετε χωρίς κανένα είδους προσωπικοποίηση δεδομένα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συγκεκριμένα τμήματα πληθυσμού. Ίσως θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω στις εποχές που δεν υπήρχε δυνατότητα να έχουμε αυτού την παρακολούθηση, το tracking, αλλά ήταν ε, δυνατό να έχουμε στοχευμένο κοινό. Δεν θα αναφερθώ στα δικαιώματα των καταναλωτών, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει και δεν θέλω να επαναλάβω τη συζήτηση, αλλά θέλω να ρωτήσω. να έχουμε συναντήσεις που θα διερκέσουν περισσότερο γιατί ήταν τόσο πλούσια αυτή, αυτές οι παρουσιάσεις και έχουμε πάρα πολλά σημεία που πρέπει να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε περαιτέρω. Έχετε νομίζω κάποιο χρόνο και στο τέλος. Νομίζω ότι θα παραμείνουν οι συνάδελφοι και εγώ συμφωνώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το πάνελ. Κύριε Μπόνη, συγγνώμη που σας περιορίζω δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να σεβαστώ το χρόνο. Η γενική εικόνα είναι, μετά τις παρουσιάσεις σας, η εξή αφενός. Έχουμε το tracking, την παρακολούθηση. Και δεν θέλουμε να παρακολουθούμαστε. Και από την άλλη, ε, είναι, έχουμε το θέμα της επιλογής και κάποιες τεχνικές δυνατότητες να αποφύγουμε την παρακολούθηση. Και παρουσιάσατε πολλές τεχνικές λύσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι εντελώς διαφορετική. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε σωστά αυτή την νομοθεσία, θα πρέπει να φανταστούμε και να δώσουμε χρόνο στις επιχειρήσεις να προετοιμάσουν κάποιες νέες τεχνικές λύσεις. Είναι δυνατό να μπει σε εφαρμογή και να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις ταυτόχρονα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, γιατί ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες έχουμε πρόβλημα με την εφαρμογή του GDPR. Και αν ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε σωστά τον κανονισμό e-privacy. Εγώ φαινώς θέλω να υπάρχει αυτός ο κανονισμός, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι πάρα πολλές λύσεις θα σχετίζονται με κάποιες τεχνικές επιλογές. Αυτό και για να έχουμε εμείς ως χρήστες περισσότερες ρυθμίσεις, περισσότερες δυνατότητες να κάνουμε την επιλογή σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς πρέπει να εργαστούμε, γιατί συζητήσαμε με τον Μάριο και θέλουμε να κάνουμε κάποιες ε, συζητήσεις σε στρογγυλή τράπεζα για να μπούμε περισσότερες λεπτομέρειες επί των τεχνικών ζητημάτων. Και θέλουμε να εξετάσουμε διάφορε πτυχέ. Είδαμε εδώ για τη διαφήμιση σε σχέση με το ΣΕΙΠΟΤΕ. Αφενό, συμφωνώ μαζί σα, αλλά από την άλλη, μπορούμε να θέσουμε και το ερώτημα αν ε, χρειαζόμαστε στοχευμένη διαφήμιση. Γιατί αν είναι στοχευμένη διαφήμιση, Φυσικά απαιτεί πρόσβαση στα δεδομένα και επεξεργασία των δεδομένων και δημιουργία προφίλ. Έτσι λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά όλες αυτές τις πτυχές για να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ε, ένας από τους προηγούμενους ομιλητές ε, είπε ότι θα πρέπει ε, να υπάρχουν πιο αυστηροί περιορισμοί στα ISP διότι μπορούν να δουν τα πάντα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Επίσης, ε, με, μου είναι δύσκολο όταν ε, συζητάμε για είναι ε, ισότιμη με τη συμμετοχή, διότι αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να αγωνίζεται σχετικά με το πώς θα έχει μια καλύτερη θέση σε αυτό. Δεν έχω πιστεί για τα ότι τι, ότι εκεί υπάρχει ισότιμη συμμετοχή με τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες, διότι έχουμε υποδομές, έχουμε υποστήριξη, όμως παρόλα αυτά οι επιφυγείς υπηρεσίες, τα OTT κατάφεραν να μπουν στι αγορέ διότι προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίε και έχουν την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών και επειδή έχουν, ε, και αυτό γίνεται επειδή έχουν στοχευμένες διαφημίσεις ε, διότι είναι καλύτερες σε όλη αυτή την πρόταση λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε να μην κινηθούμε προς τα πίσω. Υπάρχει λόγος που υπάρχουν, είναι καλά ε, και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των ε, ομιλητών. Επίσης δεν έχω ακούσει αρκετά ακόμα σχετικά ε, με την ενίσχυση των ίδιων των καταναλωτών. Αν δεν θέλουν ναι, να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μας, ας μην χρησιμοποιούμε αυτή την υπηρεσία. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Ο κύριος Αλβέχτη ε, θα προσθέσω πάνω σε αυτό, διότι αυτό και το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι ένας νόμος ο οποίος απαγορεύει ε, τον οποιοδήποτε ε, να ε, δώσει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάποιον άλλον, αλλά είναι ένας κανονισμός ή νόμος που δίνει τη δυνατότητα στους πάντες να αποφασίσουν αν θέλουν να δώσουν τα δεδομένα τους ή όχι. Και αυτό είναι στο επίκεντρο της κατανόησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που συζητάμε εδώ πέρα. Μερικές φορές λοιπόν έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν καταλάβει όλοι μας ε, ότι το να έχουμε θεμελιώδη δικαιώματα ε, και συνταγματικά πλαίσια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει με νόμους, αλλά μπορεί να αλλάχθει μονάχα να αλλάξουμε συντάγματα, συνθήκες ε, και χάρτες. Ε, στο άρθρο 8 λοιπόν της ε, χάρτας ορίζεται ξεκάθαρα ότι μπορούμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μονάχα αν υπάρχει έγκριση του προσώπου ή αν υπάρχει νόμος ο οποίος επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πλαίσιο ε, να στείλουμε κάποιον να εκπροσωπήσει μια εταιρεία ή ακόμα και έναν ολόκληρο κλάδο ε, για να δηλώσει ότι η έγκριση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ισούται ε, με αντισυνταγματικό. Δεν ξέρω, όμως θα έλεγα ότι μερικές φορές θα πρέπει να παραμένουμε κοντά ε, στα όσα συζητάμε σχετικά με τη βάση της κοινωνίας μας η οποία βασίζεται στην αυτονομία του προσώπου το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα χειριστεί ένα ζήτημα ή όχι, αν θα υπογράψει ένα συμβόλιο, αν θα δώσει δεδομένα ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να, να δίνουν αυτή την έγκριση παρά να τους αφαιρούμε αυτή την απόφαση και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό ε, και που θα ήθελα να τονίσω και επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε στο να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του προσώπου αλλά και τον ελεγκτή σχετικά με την απόφαση του αν θα δώσει τα δεδομένα ή όχι και ε, πώς η έγκριση αυτή ε, θα γίνει με έναν ε, φυσιολογικό τρόπο και όχι κουραστικό για τους πάντες. Και κάτι τελευταίο. Ο λόγος ε, για τον οποίο σε αυτό το τομέα επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα μέρη είναι επειδή δεν γνωρίζω όλα αυτά τα μέρη ε, και αν επιστρέψουμε στην βάση της οικονομία της αγοράς που αφορά την αυτονομία, συνήθως γνωρίζω τον άλλον με τον οποίο κάνω μια επιχείρηση. Όμως ε, στην περίπτωση των cookies ε, που χειρίζονται τρίτα μέρη τα cookies αυτά, δεν γνωρίζω αυτά τα τρίτα μέρη, οπότε είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια, μια σχέση για μια ενημερωμένη επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε ε, Μπόνιαν, συμφωνείτε. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ε, να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και να υπάρχει πληροφόρηση ε, προς τους χρήστες. Σεβόμενοι τις συνταγματικές υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε τώρα στην κυρία Κοπίνη. Θα μιλήσω στα ρουμάνικα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το πάνελ αυτό που ακούσαμε έχει διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους διότι κάποιος είπε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, πολύ ωραία, και είπε ξεκάθαρα ότι από την δικιά του άποψη ο γενικός κανονισμός ε, δεν φτάνει, δεν αρκεί. Συμφωνώ. Από την άλλη όμως, κάποιος άλλος προηγούμενος είπε ότι θα έπρεπε εγώ λέω ότι δεν πρέπει να λέμε θα έπρεπε, πρέπει να λέμε πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν, μιλάμε για την προστασία των καταναλωτών. Φυσικά και ο καθένας αποφασίζει μόνος του. Εγώ θέλω να ξέρω τι θα γίνει με τα δεδομένα μου, γιατί αν δεν ξέρω τι θα συμβεί με τα δεδομένα μου, πώς να αποφασίσω Μπορεί να μου έρθουν ένα σωρό διαφημίσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο χωρί να ξέρω που βρήκανε τη διευθυνσή μου. Τα ξέρω μέχρι και τι έχω φάει. Δεν υπάρχουν δηλαδή προδιαγραφέ συγκεκριμένε για τη χρήση των δεδομένων. Εγώ θέλω να ξέρω και πρέπει να είναι γνωστέ και νομικέ συνέπειε. Τι γίνεται αν κάποιο χρησιμοποιεί τα δεδομένα μου χωρίς εγώ να έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου. Μπορώ να συμφωνήσω να δώσω τα προσωπικά μου δεδομένα. Αλλά μπορεί και όχι. Αν ένα τρίτο μέρος τα χρησιμοποιήσει χωρίς τη δικιά μου συγκατάθεση, αυτό πρέπει να λύνεται. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, πάνω σε αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και χαίρομαι που η συγγήτρια ζήτησε μια συζήτηση περισσότερο σε βάθος, εκτενέστερη. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρμοδιότητα και να προστατεύεται το απόρριτο των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε Όλοι χρειαζόμαστε κάποια εγγύηση για το απόρριτο των επικοινωνιών μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, περνάμε στο πάνελ τώρα. Περιοριστείτε, οι ερωτήσεις βέβαια είναι πάρα πολύ πλούσιες αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δύο-τρία λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Μουνιώθ Μάρκος πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, Αν τα δεδομένα ε, δεν ε, μπορούν να ταυτοποιηθούν ποιανού είναι ή αυτό γίνεται σε ένα επόμενο στάδιο, τότε πρέπει να είναι προσωπικά δεδομένα από την αρχή. Σε μερικές περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι στα χέρια κάποιου τρίτου μέρους. Κανονικά αυτό που επεξεργάζεται τα δεδομένα πρέπει από την αρχή να ξέρει ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Για την νομική βάση είναι είτε για τη συλλογή, είτε για την επεξεργασία, είτε στη συνέχεια για το πού θα πάνε. Όντω πρέπει και για τα τρία στάδια να υπάρχει νομική βάση, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση από τι τρει. Μπορούμε να έχουμε μία για τη συλλογή, μία για την επεξεργασία και μία για την απόδοση των δεδομένων. Τώρα για την διάκριση ευαίσθητα, μη ευαίσθητα δεδομένα. Ναι, είναι βέβαια ένας ιδιαίτερα περίπλοκος τεχνικά κόσμος. Τα δεδομένα μπορεί να είναι στάνταρτ σε κάποιες περιπτώσεις, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγούν αυτά σε ευαίσθητα δεδομένα. Έχει να κάνει με θέματα υγείας στο οποίο μπορεί να οδηγούσουν αυτά τα δεδομένα, πληροφορίες για την υγεία του ατόμου. Οπότε πρέπει να δούμε περισσότερο το θέμα της ευαισθησίας στην επεξεργασία των δεδομένων παρά στα ίδια τα δεδομένα. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Σίγουρα χρειαζόμαστε εργαλεία για τη διαφάνεια και τον έλεγχο που θα εξελιχθούν με διαφορετικό τρόπο. Ένας χρήστης πρέπει να είναι πληροφορημένος και να μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο θέλει ή δεν θέλει την συγκεκριμένη επεξεργασία. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Όλες οι σελίδες δεν έχουν το ίδιο παράθυρο πρόσβασης στον ε, καταναλωτή, αλλά πρέπει να δίνουν πρόσβαση στον κόσμο να αποφασίζει για τα δεδομένα του και για την επεξεργασία τις οποίες θα τύχουν τα δεδομένα του. Αυτό είναι η διαφάνεια και ο έλεγχος. Οι διάφοροι φορείς Telecom μπορούν να τα δουν αυτά. Χρησιμοποιούν ε, όχι το περιεχόμενο των δεδομένων, αλλά τα μεταδεδομένα πιο πολύ. Έχουν τρόπους για να κάνουν το routing και να υπάρχει πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ευχαριστούμε κύριο Γκρούντελ. Ευχαριστώ. Να επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν, γιατί χρειαζόμαστε στοχοποιημένη διαφήμιση και προσωποποίηση. Για πολλά χρόνια ο κλάδος ε, χρηματοδοτείται από την διαφήμιση. Η απάντηση είναι ότι είχαμε μεγάλη αναλυγή από τα αναλογικά στα ψηφιακά μίντια, στα αναλογικά μέσα. Η διαφορά ήταν καταρχήν ο κατάλογος και ο χώρος ήταν περιορισμένα και όσοι επιβίωσαν σε αυτή την αναλογική κατάσταση είχαν πάρα πολύ ισχυρή θέση στην τοπική αγορά. Και γι' αυτό μπόρεσαν να πληρώνονται ακριβά για τη διαφήμιση. Τώρα στα ψηφιακά μέσα ο κατάλογος είναι πάνω κάτω άπειρος. Η αξία δεν είναι εντός του χώρου, αλλά βρίσκεται στα δεδομένα. Και αν δείτε τη διαφορά τιμών ε, μιας ε, διαφήμισης με δεδομένα που είναι στοχευμένα και προσωποποιημένα και μία χωρίς, ε, βλέπουμε πολύ μεγάλη απόσταση, είναι πολλές φορές ακριβότερη, πολύ ακριβότερη γιατί είναι πολύ καλύτερη. Μπορείτε να με εμπιστευτείτε, οι παγκόσμιοι παίκτες θα έχουν στοχευμένη διαφήμιση και θα είναι φυσικά πολύ πιο ακριβή. Αν δεν το υιοθετήσουμε δηλαδή αυτό, δεν θα μπορέσουμε κι εμείς να ανταγωνιστούμε. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τους ε, καταναλωτές και την ανδυναμωσή τους. Ε, ναι, σας έδειξα το εργαλείο μας πριν. Όμως αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα είναι ε, να δείξουμε ποια δεδομένα έχουμε για σένα και για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιήσουμε και τι μπορείς να κάνεις να μας σταματήσεις αν θέλεις ή αν θες να μας το επιτρέψεις να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει με διαφανή τρόπο. Το γεγονό είναι ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε από κοινού με του πελάτε μα. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε αυτό στου παγκόσμιου παίκτε που θα το κάνουν αντίμον. Και αυτό θα συνέβαινε αν θα το έκαναν οι φιλομετρητέ οι browser. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χιτφέκη. Για να μην επαναληφθώ, θα επικεντρωθώ μόνο σε λίγα σημεία. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι βρίσκω κάπως προσκλητικό να θεωρεί κανείς τη διαφήμιση ως τον ακρογωνιό λίθιο των ε, δωρεάν μέσων ε, και δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό ο χαρακτηρισμό του προβλήματος και σίγουρα η προστασία του απορρίτου δεν θέτει σε κίνδυνο την ε, ανεξαρτησία των μέσων. Τώρα, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και την επιβολή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω χρόνος Τώρα έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή γιατί είχαμε ε, ουσιαστικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα κτλ. Νομίζω ότι λύθηκε αυτό από το ΕΠΡΑΒΕΣΙ και από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Για τους χρήστες και την προσαρμογή τους στην πραγματικότητα, θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και να αναλάβουν τον έλεγχο οι χρήστες. Ίσως αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι να ευαισθητοποιήσουν περισσότερα γιατί βλέπουμε ότι έρχονται άνθρωποι να παραπονεθούν σε εμά, αλλά αν και δεν το έκαναν, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν και ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο, μπορεί να μην καταλαβαίνουν ποια είναι η εικόνα. τώρα αυτό που μας δείχνουν οι διάφορες παράμετροι είναι ότι θέλουν υψηλότερα πρότυπα και θέλω να ε, σας ε, ε, κάνω και μια έκκληση σε σχέση με το θέμα του όρου χρήστη και του καταναλωτή, του όρου καταναλωτή, γιατί δεν σχετίζονται με αυτή τη σχέση ε, ουσιαστικά και τα δύο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συλλογή και τη χρήση, είναι προφανώς ότι και τα δύο καλύπτονται, αλλά συμφωνώ ότι ο κανονισμός η privacy θα πρέπει να βελτιωθεί για την πτυχή που σχετίζεται περισσότερο με, την, ε, με το στάδιο του χρήστη. Ξέρω ότι θα θέλατε να πείτε παραπάνω. Και τέλος ο καθηγητής. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Μπόνι για το τι θα πρέπει να έχουμε θεσπίσει πριν έχουμε μια οδηγία η privacy και το να αναπτύξουμε τις σχετικές τεχνολογίες, τις αναπτύσσουμε αυτές εδώ και 20 χρόνια και μαζί με τη βιομηχανία και αυτό που βλέπουμε πάντα, κυρίως από τέρους από τον κλάδο και από τη βιομηχανία, παντού είναι ότι αν έχουμε σαφή κανονισμό για το τι μπορούμε να κάνουμε και το τι πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι και να φτιάξουμε καλά πράγματα. Αν είναι σαφής ο κανονισμός, τότε έρχονται οι μεγάλοι και κόβουν τον προπολογισμό μας ε, για τα καλύτερα πράγματα. Αυτό γίνει με την ιδιωτικότητα, λιγότερο με την ασφάλεια, αλλά γίνεται ακόμη και αν ε, συγκρίνει τον προπολογισμό για την ιδιωτικότητα και για την ασφάλεια, ε, βλέπουμε, παίρνουμε το σχάρι πόσα χρήματα πηγαίνουν στο ένα και πόσα πηγαίνουν στο άλλο. Έτσι λοιπόν, χρειαζόμαστε σαφή δήλωση από τους νομοθέτες ε, έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν με αυτό το θέμα και οι ενδιαφερόμενοι. Τώρα, για τους καταναλωτές, κατά πόσο πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Τους εμπιστευόμαστε, όμως το θέμα είναι ουσιαστικά ε, τι σημαίνει το να έχουμε ιδιωτικότητα. Ε, είναι σαν να πλένει κανείς τα δόντια του. Πρέπει να αφιερώσει χρόνο, Όμω, ε, μόνο μακροπρόθεσμα θα έχει αποτελέσματα ο σεβασμό τη ιδιωτικότητα ε, και ουσιαστικό το ίδιο γίνεται σαν να πηγαίνει ε, στη βιομηχανία γλυκών και να ε, ρωτάς αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα γλυκά. Όμως έχουμε αναπτύξει μία έννοια για την ενημέρωση των πολιτών, ε, για τις ε, μεταφορές ε, των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας, γιατί οι περισσότεροι στο διαδίκτυο ε, μας λένε από κάτω «Α, έχεις διαβάσει τους όρους». Κανένας, τέλος πάντων, δεν μπαίνει στον κόπο να τα διαβάσει όλα αυτά, απλά κάνει ένα κλικ στο «Ναι». ουσιαστικά ε, υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα ε, τα οποία αναπτύχθηκαν ε, από τις υπηρεσίες οτιτής. Αυτό όμως τώρα τι σημαίνει ότι δεν θέλει η Google ούτε όσοι προσφέρουν υπηρεσίες οτιτή να τα δώσουν αυτά. Θέλουν να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους. Δεν θέλουν να ενημερώνονται οι καταναλωτές. Αν ε, βέβαια παράσχαμε τις πληροφορίες θα μπορούσαμε να είμαστε σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Ε, τώρα δεν ξέρω αν κατάλαβα πολύ καλά την ε, ερώτησή σας. Τι είπατε, ε, ουσιαστικά αναφερθήκατε στην προσωποποίηση των δεδομένων, ε, αν κάποιος πάρει ε, προσωπικά δεδομένα και τα επεξεργαστεί, για να δούμε αν εξακολουθούν να είναι προσωπικά αυτά τα δεδομένα, νομίζω πρέπει να το ψάξουμε περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας σήμερα. Σας παρακαλώ να μείνετε σε επαφή μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για τις οπτικές που μας παρουσιάσατε εδώ. Περνάμε τώρα ε, στην τρίτη συνεδρίαση. Θα παρακολουθήσω λοιπόν τους ε, συναδέλφους να ανέβουν στο Προεδρείο. Θα σας ε, παρουσιάσω καθώς έρχεστε. Θα εξετάσουμε σε αυτή την τρίτη συνεδρίαση την ε, εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των επικοινωνιών. Όταν ε, τη θέση τους οι ομιλητές θα ξεκινήσουν κατευθείαν. Um, Συνάδελφοι, αυτοί ε, που θα μείνουν, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την τρίτη συνεδρίαση. Ε, όπως ε, πάντα, στην τελευταία συνεδρίαση ε, οι ομιλητές έχουν πίεση χρόνου και γι' αυτό το λόγο θα είμαι λίγο πιο αυστηρός με το χρόνο και ε, θα ήθελα ε, να σας ζητήσω άμα μπορείτε, να περιοριστείτε σε 7 λεπτά ώστε να μας απομείνει χρόνος για τον γύρο των ερωτήσεων. Ο πρώτος ομιλητός ε, λοιπόν είναι ο κύριος ε, Ηλίας Χατζός ε, από την σύματα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την άποψη της βιομηχανίας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, εκπροσώπη του ε, Συμβουλίου της ε, Επιτροπής ε, των Κρατών Μελών, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τους διοργανωτές που μου έδωσαν τη δυνατότητα να βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να επικεντρωθώ σε ζητήματα τα οποία αφορούν ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλεια που, είναι, που αποτελούν τους βασικούς στόχους της συγκεκριμένης οδηγίας. Έτσι λοιπόν το ερώτημα είναι αν το e-privacy υπηρετεί ε, έναν ε, ε, στόχο δημόσιας πολιτικής. Έχουμε, έχουμε τις πληροφορίες που καλύπτονται από το Γενικό Κατελληνισμό, έχουμε τις υποδομές που καλύπτονται από την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, έχουμε τις ταυτότητες που καλύπτονται από το AIDAS, τι γίνεται όμως με τις επικοινωνίες εκεί. Έχουμε, αν δεν επιθυμούμε εμπιστευτικότητα, εκεί υπάρχει ένα σημαντικός ρόλος ε, να παιχθεί, όμως για να γίνει αποτελεσματικός θα πρέπει να είναι ε, σωστά στοχευμένος ε, και να συμφωνεί με άλλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε επανειλημμένα αρκετά ε, για τις επιφυείς υπηρεσίες, ε, για, την επίρρηση, για τις ε, επιρροές που έχουν αλλά και άλλους τομείς της βιομηχανίας που επηρεάζονται από την οδηγία. Όμως κάτι το οποίο στοχεύει είναι το Internet of Things, το Internet των πραγμάτων, ε, της ε, επικοινωνίας και την ασφάλεια. Είναι αναγκαίο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι το ακούσαμε από αρκετούς ειδικού ε, σε ζητήματα ασφάλεια τις τελευταίες εβδομάδες το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να προστατεύουμε τη μηχανή προς μηχανή επικοινωνία στο ίντερνετ των πραγμάτων. Όσον αφορά εμένα λοιπόν η διαφάνεια αλλά και η ασφάλεια είναι σημαντικά χαρακτηριστικά προϊόντων ποιότητας. Εκτός λοιπόν από την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια τα οποία συζητώνται θα πρέπει να υπάρχει και το ζήτημα της ταυτοποίησης, της πιστοποίησης και όλα αυτά είναι πράγματα πάνω στα οποία εργάζεται η IoT. Όλα αυτά λοιπόν έχουν κάθε λογική η ιδέα όσον αφορά τη συζήτηση για τους ε, φιλομετρητές και τα cookies ε, έχει λογική κατά τη γνώμη μας. Ε, η διάταξη σχετικά με τα cookies δεν είναι αποτελεσματική διότι βλέπουμε οι χρήστες απλά να κρυκάρουν accept, αποδοχή Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόκληση εδώ πέρα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε ε, ένα ε, πλαίσιο, έναν ελεγκτή πύλη, όπου θα αναγκάσουμε ε, τους πολίτες να επικεντρώνονται και τους χρήστες να επικεντρώνονται σε ένα μονάχα σημείο. Η ιντερνετική πρόσβαση λοιπόν, η διαδικτυακή πρόσβαση γίνεται ε, ανεξάρτητη της χρήσης φιλομετρητών. Έτσι λοιπόν όλη η συζήτηση του πρώτου μέλους ε, και τρίτου μέλους μπορεί να είναι προβληματική διότι ε, όταν χρησιμοποιούμε φιλομετρητή είναι καλύτερο, το πρώτο μέλος είναι καλύτερο και έτσι λοιπόν όλα τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να δώσουν την συγκατάθεση. Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ποιοι τομεί χρειάζονται βελτίωση λοιπόν στο e-privacy. Έχουμε δει λοιπόν μια ξεκάθαρη αποδοχή της ε, διαχείρισης ε, και της επεξεργασίας ε, δεδομένων για ζητήματα κυβερνού ασφάλειας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συγχαρούμε την Κομισιόν που κάνει το συγκεκριμένο βήμα και αναγνωρίζει την ε, σημασία της κυβερνοασφάλειας τη ηλεκτρονικές επικοινωνία. Αν όμως το δούμε από πλευράς κατηγοροποίησης, νομίζω ότι η Κομισιόν ε, το προσέγγισε ορθά με την έννοια ότι θα πρέπει να προστατεύουμε τα μεταδεδομένα και ε, τα περιεχόμενα, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά για την παροχή σωστή προστασία. Η εξαίρεση λοιπόν είναι σωστή. Η ε, ο κατακαιρματισμός δεδομένων είναι ορθός, όμως το εύρος της εξαίρεσης είναι λάθος. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γραφεί η εξαίρεση και συγκρούεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων είναι ότι με βάση ε, το, ε, το e-privacy, η πρόσβαση υπάρχει μονάχα για τα OTT και τα telecoms όμως η πρόσβαση στα δεδομένα για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν ε, κάθε συμφέρον όμως ο υπάροχη προστασίας ή ε, μια τράπεζα ε, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα αφύσικο αποτέλεσμα λόγω του ότι επικεντρωνόμαστε στο εύρος ε, του e-privacy με αποτέλεσμα να έχουμε ένα διεστραμμένο αποτέλεσμα δίνουμε τα κίνητρα σε όλους όσους βασίζονται στον γενικό κανονισμό να χρησιμοποιούν την επεξεργασία δεδομένων για ζητήματα ασφαλείας ε, και να το κάνουν σε πιο έντονο βαθμό, όπως είναι για παράδειγμα η ε, διεύθυνση IP ενός υπολογιστή με ιό. Ε, ή το URL ε, που χρησιμοποιείται για phishing, όλα αυτά δεν περιλαμβάνονται ε, στο, στην τωρινή πρόταση. Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ευθυγράμμιση με τον γενικό κανονισμό αλλά και με, την, με το e-privacy. Επίσης λοιπόν για να ξεκαθαρίσω αυτό που θέλω να πω, δεν φαίνεται ίσως καθαρά στη διαφάνεια, διαφάνεια άμα εξετάσουμε την ε, οδηγία του 2009 ε, εκεί δίνει πρόσβαση ε, σε παρόχους τεχνολογικής ασφάλειας. Ο γενικός κανονισμός ε, δίνει την ίδια δυνατότητα σε ε, ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και σε ε, παρόχους τεχνολογικής προστασίας, όμως πλέον στο νέο κανονισμό αυτό περιορίζεται μονάχα στις επιφυγείς υπηρεσίες. Για άλλη μία φορά λοιπόν, ιστορικά, τόσο το 2009 όσο και ο Γενικός Κανονισμός ε, έχουμε κείμενα τα οποία είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου ε, για την κυβερνοασφάλεια, για την ε, προστασία των ψηφοφόρων σας, των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν αυτό που σας λέω όπως κάνατε δύο φορές στο παρελθόν ξανακάντε το, διορθώστε το κείμενο θα μπορούσαν οι διατάξεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας να βελτιωθούν και πιστεύουμε πως ναι. Αρχικά υπάρχει η σωστή στόχευση, όμως υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Ε, για εμάς λοιπόν το ζήτημα είναι να ε, παραδώσουμε δυνατότητες ασφάλειας ε, σε αντίθεση με το να δώσουμε απλά την υποχρέωση, να ορίσουμε την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και αυτό βασίζεται στην εμπειρία μας με βάση το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων το οποίο το βλέπουμε ε, ιδιαίτερα συχνά εξαιτία αυτού. Επίσης, ε, απαιτείται ε, στο πλαίσιο της ασφάλειας πρόσβαση στο τελικό σημείο και το άρθρο 17, αν θα πρέπει να ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης, Εμεί δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μερικά σχόλια ακόμα εντάχει. Ε, δεν είναι ε, μία σκέψη που σχετίζεται με την ασφάλεια, αλλά αφορά το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργούμε. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό υπάρχει ένας, ένα πλαίσιο σχετικά με την πρόσβαση των δεδομένων για ολόκληρη την ε, κοινότητα. Εσείς έχετε να λάβετε μία απόφαση και όσο πιο ε, αποκλειστική κάνετε αυτή την πρόσβαση, τόσο πιο ε, δύσκολο θα είναι να έχουμε ένα οικοσύστημα, ένα πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας και θέσεων εργασίας που επιζητάτε και ε, το ζήτημα της ε, πρόσβασης ε, για την αστυνομία καλύπτεται στο e-privacy, είναι σωστό να περιλαμβάνεται, όμως επειδή η εξαίρεση είναι πολύ ανοιχτή για τα κράτη-μέλη, θεωρούμε ότι θα πρέπει να, να το ορίσουμε καλύτερα με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τώρα έχουμε τον κύριο Γκουλιέρμο Πέλτρα, ε, ο οποίος θα ε, μιλήσει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε την ΠΕΚ που είναι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό τον οποίων εκπροσωπούνται 31 χώρε με του αντίστοιχου οργανισμού προστασία των καταναλωτών. Ήρθαμε να προσφέρουμε και εμεί τι απόψει μα για αυτό το τόσο σημαντικό σχέδιο νομοθεσία που προτείνεται. θεωρούμε πολύ καλό σημείο κίνηση στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συζήτηση και να γνωρίζουμε την προσπάθεια της Κομισιόν μετά από μεγάλη πίεση που υπήρξε για την νομοθεσία αυτή. Από όσα ακούσαμε και από τα προηγούμενα πάνελ πρέπει να υπενθυμίσουμε γιατί έχουμε και γιατί είναι τόσο αναγκαία αυτή η νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα, όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ο επόπτης δεδομένων είπε νωρίτερα, είναι θέμα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιωτικού βίου. Άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όπως ε, και η οδηγία για την ή ε, Protection, έτσι και ο κανονισμός τώρα θα αποτελεί ένα συμπλήρωμα, ένα επιπλέον στρώμα προστασίας του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Επιπλέον, θα σκεφτούμε, ο κανονισμός μπορεί να αποτελέσει έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα σε ένα φιλικό πλαίσιο ανταγωνισμού και μπορεί να βοηθήσει και με καινοτομία με τη ε, δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών προς το συμφέρον του καταναλωτή. Υπάρχουν δηλαδή πολύ καλοί λόγοι για, τον, για τους οποίους ο κανονισμός αυτός εξυπηρετεί. Αναλύοντας την πρόταση και βάσει και όσων είπε και ο κύριο Άλμπρεχτ νωρίτερα, υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να αλλάξουν. Εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα κάποιε σκέψει μου για το πόσο οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν. Πρώτον, η σημασία του απόρριτου των επικοινωνιών. Ακούσαμε σήμερα ότι αυτό είναι ο τρόπο για να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών. Η κυρία Σπανού σήμερα είπε ότι 92% των καταναλωτών που έχουν ερωτηθεί θέλουν να προστατεύεται το απόρριτο. Η πρόταση αυτή λοιπόν επεκτείνεται για να καλυφθούν όλες οι υπηρεσίες επικοινωνιών, όχι μόνο οι παραδοσιακές. Και οι over the top, όπως λέγονται, οι OTT. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι καταναλωτές θέλουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Ό,τι υπηρεσίε όμως και αν χρησιμοποιούν. Ένα σημαντικό θέμα που σημείωσε κάποιος νωρίτερα και θέλω να το επαναλάβω κι εγώ είναι ότι μιλάμε και για αποθηκευμένα δεδομένα τηλεπικοινωνιών. Κάτι άλλο σημαντικό που έχει να κάνει με τον κανονισμό αυτό και που πρέπει να διασφαλίσει ο κανονισμός είναι η ασφάλεια των δεδομένων. Εδώ πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση του κανονισμού αυτού με τον προτινόμενο κώδικα επικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που περιλαμβάνει σημαντικά άρθρα για την ασφάλεια. Άρα πρέπει να θυμόμαστε την σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά μέσα. Ακούσαμε τον συνάδελφο πριν από λίγο από τη Σίμαν που μιλάει για την ασφάλεια και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Ακούμε ανησυχητικά νέα για το πώς ε, κλέβονται δεδομένα, πως ακόμα και τα παιχνίδια μπορούν να κατασκοπευτούν και να μπορεί κανείς με τον τρόπο αυτό να κλέψει δεδομένα. Έχουμε μια εκστρατεία εμείς για ένα παιχνίδι που όντως κλέβονται δεδομένα από αυτό, μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει για να πάρει πληροφορίες και στη συνέχεια να τις μεταφέρει σε τρίτα μέρη. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι εδώ προστατεύουμε το κοινό ό,τι θέλουμε για τα παιδιά μας, αλλά όχι μόνο για τα παιδιά μας, για όλους μας. Ένα σημαντικό στοιχείο επίση είναι ότι ο κανονισμός για το e-privacy δεν πρέπει να περιορίζει τις δυνατότητε του καταναλωτών να προστατευτούν με νέες τεχνολογίες όπως είναι η κρυπτογράφηση. Κάτι άλλο, επίση σημαντικό, πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον και πώς θα προστατευτεί το θέμα αυτό και στο μέλλον από τον ετοπισμό και την παρακολούθηση. Είπαμε ότι θέλουν εξορισμού την προστασία οι καταναλωτές όταν χρησιμοποιούν κάποιο φιλομετρητή. Αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση κανονισμού, ενώ δεν υπάρχει τώρα. Όπως είπε νωρίτερα και ο κύριος Μποργέζιους και το βλέπουμε αυτό και στην γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας για το άρθρο 29, η προστασία του ιδιωτικού βίου εξορισμού δεν είναι το ίδιο με την επιλογή εξορισμού. Πρέπει να είναι ο κανόνα. Και δεν μιλάμε μόνο εδώ για τους φιλομετρητές, πρέπει να μιλήσουμε και για άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας που επιτρέπουν στους καταναλωτές να επικοινωνούν μεταξύ τους ή με μηχανήματα, είτε συστήματα λειτουργίας ε, των ε, κινητών, είτε εφαρμογέ κλπ. Ένα σημαντικό άρθρο στην πρόταση αυτή είναι το άρθρο 8, το οποίο αναφέρεται στην ε, προστασία των μηχανημάτων. Και Κοιτάξτε, σε αυτό το μηχάνημα υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα ιδιωτικού βίου μέσα σε αυτό το μηχάνημα από ό,τι έχω σε ολόκληρο το σπίτι μου. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι έχουμε προστατευτικά μέτρα για τα μηχανήματα αυτά, είναι ζωτική σημασία περισσότερο από ποτέ σήμερα. Το άρθρο, λοιπόν, το άρθρο αυτό επίσης πρέπει να προβλέψει και το μέλλον. Δεν μιλάμε μόνο για τα cookies εδώ, υπάρχει το 8 8.2β που είπαμε ε, για τον εντοπισμό, την παρακολουθούση που δεν πρέπει να γίνεται χωρί ε, συνένεση. Πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα αποφεύγει επίσης τον κατακλυσμό από αιτήματα για συνένεση. Το άκουσα από πολλού σήμερα, οπότε πρέπει και εγώ να πω εδώ ότι πρέπει να σκεφτούμε τα θετικά της ιδέας του κατά πόσο πρέπει να επιτρέψουμε ή όχι τα λεγόμενα tracking walls. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τζουζέ Πεντακίστο ο οποίος προέρχεται από την Εθνική Αρχή Προστασία των Δεδομένων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να σας θέσω μια ερώτηση θα, δέχεσταν, θα δέχόσασταν οι προσωπικές σας επικοινωνίες ε, να δημοσιεύονταν σε όλους και να παρουσιάζονται στην τηλεόραση απόψε. Αν απαντήσετε όχι, όπως φαντάζομαι, μπορείτε να καταλάβετε εύκολα τη σημασία της εμπιστευτικότητας του απορρίτου. Είναι ε, κάτι που ε, ουσιαστικά αφορά τον ενδόμηχο κόσμο μας, αλλά είναι και κοινωνική αξία. Χωρίς ε, το απορρίτο δεν θα είχαμε τηλεπικοινωνίες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ειδικού κανόνες ε, πέρα από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων. Πρέπει να προστατεύσουμε το απόρριτο και την ιδιωτική ζωή και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Γιατί κανονισμό. Η τεχνολογία είναι το κλειδί για την απάντηση. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται εμπόρευμα. Όσο μειώνεται το κόστος, τόσο η επεξεργασία των δεδομένων ε, απομακρύνεται από την Ευρώπη και από τα άτομα προς ε, ένα μικρό αριθμό πολύ αποτελεσματικών παγκοσμίων παικτών. Σήμερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ε, διάφορες εφαρμογές φωνής, βίντεο και αποστολής μηνυμάτων με έναν απρόσκοπτο τρόπο και αναμένουν το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας. Ε, νομίζω ότι ο κανονισμός είναι ένας, ε, ο καλύτερος μάλλον, ε, η καλύτερη επιλογή για να δώσουμε μία νέα εξισορρόπηση στα αποτελέσματα αυτής της εμπορευματικοποίησης. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα με μια γενική απαγόρευση για την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός αν έχουμε κάποιες εξαιρέσεις. Καταρχήν, την αναγκαιότητα των δεδομένων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ε, ανωνυμοποίηση των δεδομένων και την συνένεση των χρηστών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι επαρκέ για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι όσο πιο εναρμονισμένο και να ισχύει για όλα τα είδη ε, δεδομένων ε, και περιεχομένου και μεταδεδομένων και σε όλα τα είδη επικοινωνιών. Τώρα να αναφερθώ στο θέμα των ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Η ανωνυμοποίηση είχε ήδη εισαχθεί ως επιλογή στην οδηγία ως εναλλακτική στη διαγραφή των δεδομένων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Η πρόταση θέτει την ανομοποίηση στην ε, αρχή του κύκλου της ζωής των δεδομένων και προσφέρει μία διπλή ζωή στα δεδομένα. Μία ζωή ως παραδοσιακά προσωπικά δεδομένα και μια άλλη ζωή ως ανώνυμα δεδομένα που και πάλι θα προσφέρει στους αρμόδιους της επεξεργασίας τεράστιες ευκαιρίες για πολλές εφαρμογές σε ό,τι αφορά το δίκτυο των πραγμάτων και τα μαζικά δεδομένα. Στις μελλοντικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες η εφαρμογή της ανωνυμοποίησης θα απαιτεί κατά την άποψή μου τρεις μεγάλες δεσμεύσεις από τους αρμόδιους της επεξεργασίας. Καταρχήν διαφάνεια στο πεδίο ε, εφαρμογής και στη μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται για την ανομοποίηση. Δεύτερον, μία προκαταρκτική μελέτη αντικτύπου της, του απορρίτου με υποχρεωτική διαβούλευση με τις αρχές προστασίας των δεδομένων και ένα εύκολο opt-out τρίτον για τους χρήστες, ακόμη και από την ίδια την ανομοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι η ανομοποίηση η οποία θα διέπεται από κανόνες, μπορεί να γίνει πραγματική ευκαιρία ε, που θα είναι φιλική προς την ιδιωτικότητα. Η σημερινή πρόταση ε, δίνει πολύ αδύναμες υποχρεώσεις στους αρμόδιους της επεξεργασίας ε, και αφήνει ε, ουσιαστικά τη μόνη δυνατότητα του χρήστες, δεν αφήνει άλλη δυνατότητα παρά να σβήσουν τη συσκευή τους. θέλω να αναφερθώ ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη δέσμευση από τους αρμόδιους επεξεργασίας γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ασημοτρία ε, για τα μας δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεχθούν οποιαδήποτε στιγμή με πολύ μικρή παρέμβαση από τα υποκείμενα. Οι σημερινέ προτάσεις δεν επιτρέπεται για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ε, και θα έλεγα ε, ότι η εφαρμογή των λύσεων opt-out ε, που να μην είναι λύσεις ότι σβήνω τη συσκευή θα πρέπει να δίνεται και στους αρμόδιους επεξεργασίας αλλά και στους κατασκευαστές. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των αποθηκευμένων δεδομένων και σε τερματικά όπως ε, τα cookies ε, που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση οι εκδότες συνήθως ελεπιδρούν με πάρα πολλά άλλα μέρη για διάφορους σκοπούς και κάνουν την πλογήσή μας κάτι λιγότερο από εμπιστευτική οι χρήστες δεν γνωρίζουν αυτές τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις και οποιαδήποτε λύση είτε το δέχεσαι ε, είτε δεν έχεις πρόσβαση δεν είναι δίκαιη. Επίσης δεν σέβεται την απέτηση της συνένεση. Η εμπιστοσύνη στο περιβάλλον του διαδικτύου θα επωφεληθεί πάρα πολύ από την εισαγωγή μια υποχρέωση διαφάνεια καταρχήν για την ύπαρξη αυτών των ελεπιδράσεων και δεύτερον ε, σαφών τεχνικών προτύπων για την ταξινόμηση των σε ένα σκοπό. Παραδείγματο χάρη, κούκκι παρακολούθηση, κούκκι μέτρηση, ε, ε, το κρατηρίο κτλ. Σύμφωνα με την πρόταση, η συνένεση στο διαδίκτυο μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας κάποιους τρόπους που διατίθεται στους φιλομετρητές η ιδέα είναι να έχουμε κεντρική συνένεση να, μάλλον να συγκεντρώσουμε τη συνένεση σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνά. Ε, όμως δεν αρκεί να δίνουμε επιλογές για να ισχύει η συνένεση, αλλά είναι πολύ σημαντικές και οι αρχικές προϋποθέσεις και ε, ε, η διαμόρφωση ε, εξορισμού θα πρέπει να γίνεται με το πιο φιλικό τρόπο προς, την, προς το απόρριτο. Επίσης, ε, θα πρέπει ε, ουσιαστικά να έχουμε δεσμεύσει στο σερμό τη επεξεργασία, όπω ε, παραδείγματο χάρη είναι το device fingerprinting. Τώρα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την ακαιρότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Αν ε, πληροφορίε χρησιμοποιούνται για να ελέγχουμε τι συσκευέ που χρησιμοποιούν καθημερινά, σκεφτείτε τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα ή άλλε εφαρμογέ μηχανή προ μηχανή, μια γενική υποχρέωση για την ακαιρότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που εξακολουθεί να λείπει μαζί με την προστασία τη εμπιστευτικότητα μπορεί να παράγει έχει ε, μελλοντικές ε, δικλείδες ασφαλείας ε, κατά των απειλών και να προωθήσει ταυτόχρονα τη λογοδοσία και να διευκολύνει την επιβολή. Όλα αυτά τα κενά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, αν δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδίκτυο το οποίο ουσιαστικά θα διαιρεί τους πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε νέες τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες γιατί δεν θα αρκούν τα παλιά εργαλεία. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που μου έδωσε την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου για τον κανονισμό ή e privacy. Τώρα από σας εξαρτάται. Έχετε την ευθύνη να αποφασίσετε για το πώς ε, θα μοιάζει ο τρόπος που θα επικοινωνούμε στο μέλλον αυτό δεν είναι μια ξεχωριστή διάσταση των ζώων μας, είναι μια σημασία διάσταση, καθώς ε, η σφαίρα των πληροφοριών γίνεται όλο και περισσότερο η κύρια διάστασή μας ε, ως ψηφιακά ανθρώπινα όντα εμείς. Ε, θα επικοινωνούμε με εμπιστοσύνη και θα δημιουργήσουμε νέες αξίες για όλους ή θα έχουμε διενέξεις σε ό,τι αφορά ε, ουσιαστικά το χτίσιμο μιας διάβρωσης του πλούτου. Αυτή είναι η ερώτηση και σας εύχομαι κάθε σοφία που χρειάζεστε για αυτό το λεπτό καθήκον. Σε σας ήσασταν στο τέλος, ε, γιατί λυπάμαι που είστε και στο τελευταίο πάνελ, γιατί κουράζονται οι συνάδελφοι εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι όσο ένα σημείο μπορούν να αντέξουν. Βλέπω ότι κι εσείς ε, κουράζετε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνεισφορές σας ε, είναι λιγότερο πλούσιες. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Μεταδίδεστε και μέσω του διαδικτύου. Να έρθουμε τώρα στον τελευταίο μιλητή, ο κύριος Μπενζαμιστράς, μηχανικός λογισμικού από το Facebook. Stick to <laughs> παραμείνετε στα 7 λεπτά άμα γίνεται. Ε, ε, ε, όσον, ως μηχανικός λογισμικού έχω χρονομετρήσει ακριβώς την ομιλία μου και μπορώ και τη βάζω μέσα σε 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Γνωμοπάτρια, σε αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ονομάζομαι ε, Benjamin Strass ε, και είμαι ε, μηχανικός λογισμικού στο Facebook. Επικεντρώνομαι στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των χρηστών μας και θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας παρουσιάσω τις απόψεις του Facebook ε, σχετικά με το πώς ο προτινόμενος ε, ε, κανονισμός θα επηρεάσει τις υπηρεσίες. Από την εφαρμογή της οδηγίας e έχουμε δει μια αλλαγή στην φύση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας. Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν αυτές για τη μεταφορά μηνυμάτων από το σημείο α στο β, ενώ πλέον ε, απαιτούν περισσότερα. Χρησιμοποιούν ε, email τα οποία θα πρέπει να φιλτράρουν τα spam, να οργανώνουν τα inbox, ε, να έχουν ακόμα και δυνατότητα μετάφρασης το χρησιμοποιούν αυτό ακόμα και για να καλέσουν ταξί, να ε, ε, λάβουν οδηγίες. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια υπηρεσία που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ήθελα λοιπόν να σας πω πώς εμείς εργαζόμαστε για να δώσουμε τη δυνατότητα στου ανθρώπου να εκφράζονται αλλά ταυτόχρονα να μείνουν ε, συνδεδεμένοι με έναν ασφαλή τρόπο. Ε, ένα παράδειγμα θα είναι να έχουμε έναν βοηθό στο εσωτερικό του Messenger το οποίο αυτόματα θα βοηθά του χρήστε να κάνουν διάφορε δραστηριότητε ιδιότητε. Ένα άλλο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για όλου μα του ε, ε, για όλου μα του χρήστε, είναι ε, ένα προϊόν το οποίο ονομάζουμε Automatic Alternative Text, αυτόματο ενηλεκτικό κείμενο το οποίο περιγράφει το περιεχόμενο εικόνων για άτομα με προβλήματα όρασης. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω πώς το χρησιμοποιεί το Facebook αυτό μέσω ενός βίντεο.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 το συγκεκριμένο προϊόν αναπτύχθηκε ύστερα από ε, την ανάλυση περιγραφών φωτογραφιών τα οποία απεστάλησαν στο Facebook. Θέλουμε να το κάνουμε διαθέσιμο αυτό στο Messenger στο ε, μέλλον ε, και να δίνεται η δυνατότητα για όλες τις φωτογραφίες. Αυτό έχει τη δυνατότητα λοιπόν να διευκολύνουμε την επικοινωνία και να γίνεται αξιολόγηση του περιεχομένων. Και τέλος θα ήθελα να σας μιλήσω για τη δουλειά που κάνουμε σε συνεργασία με άλλους για να είναι η ε, online εμπειρία πιο ασφαλής για τους ε, χρήστες. Εκτός από ε, τις υπηρεσίες mail και messenger έχουμε τη δυνατότητα να βρεθεί malware. Για παράδειγμα έχουμε την δυνατότητα παιδικής, να εντοπίζουμε εικόνες παιδικής πορνογραφίας οι οποίες με αποτέλεσμα να κρατούμε την κοινότητά μας ασφαλή. Με αυτόν τον ε, τρόπο έχει εξελιχθεί η επικοινωνία σήμερα η οποία είναι πιο ε, έξυπνη, πιο ε, ασφαλής. Ως ε, ε μηχανικός λογισμικού επικεντρώνουμε ε, πάνω σε αυτό και ενθουσιάζουμε σε ένα αυτό, ώστε να δημιουργήσουμε νέες εμπειρίες και νέες τεχνολογίες, όμως ο προτινόμενος κανονισμός απειλεί να περιορίσει την τεχνητή νοημοσύνη διότι αντιμετωπίζει ως παράνομες αυτές τις τεχνολογίες ε, και απαιτείται έγκριση για κάθε χρήση. Ενώ εμείς στο Facebook πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι χρήστες να έχουν ε, τον έλεγχο του του τι συμβαίνει με τα δεδομένα των χρηστών και έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ε, διαφάνεια. Ε, εάν ζητάμε συνεχώς ε, την έγκριση, τότε περιορίζεται ο έλεγχος, διότι έχουμε βρει ότι εάν οι χρήστες βλέπουν ξανά και ξανά το ένα pop-up μετά το άλλο, απλά πατάν τυπικά ναι να αντιδρούν με αποτέλεσμα, να υποβιβάσουμε τις περιπτώσεις που είναι απόλυτα αναγκαίο. Δεύτερον, αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Για παράδειγμα, όσοι χρησιμοποιούν malware, σπάμε εικόνες παιδικής πορνογραφίας. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το κάνουν, ε, διότι ε, θα επιλέξουν να εξαιρεθούν ε, θα πρέπει να μιλάμε για την προστασία των υπηρεσιών και όχι την γενικότερη κοινότητα. Επίσης, οι απαιτήσει έγκρισης μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη νέων υπηρεσιών διότι το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε αντίθεση με μια άλλη ε, νομική βάση που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτών των ε, τεχνολογιών όπως είναι ε, το κείμενο που παρουσιάσαμε στο βίντεο πριν. Για όλους αυτούς τους ε, λόγους θα πρέπει να δώσουμε έμφαση ε, στην αξιολόγηση των ε, δεδομένων επικοινωνιών που, θα αποτρέπουν, που δεν θα αποτρέπουν την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως είναι το Facebook Messenger. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουν σήμερα και αδειμονώ στο διάλογο που θα ακολουθήσει σχετικά με τον προτινόμενο κανονισμό σας. Ευχαριστώ πολύ και επίσης ευχαριστούμε για το ταξίδι σας από το Σαν Φραντσίσκο για να είσαστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ευχαριστώ ολόκληρο το πάνελ για τις παρουσιάσεις σας. Και όπως κάνουμε πάντα, θα ακούσουμε ερωτήσεις, η συγγήτρια πρώτα απ' όλα και μετά οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση μου είναι για το Facebook. μια που συζητάμε και το πεδίο εφαρμογή. Πώς εσείς αντιλαμβάνεστε το Facebook. Είναι ένα δίκτυο πρόσβασης. Πώς βλέπετε εσείς να ταιριάζει με το πεδίο εφαρμογής. Ποιος είναι ο χώρος που αντιστοιχεί στο, στο facebook είναι δημόσιος, ο χώρος είναι ιδιωτικός, τι είναι. Βιβλίο, facebook. Τα προβλήματα τώρα με την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ που υπογραμμίσατε τόσο πολύ την ανάγκη να καταλάβουμε το θέμα του απόρριτου και της ασφάλειας, ότι πρόκειται για τις δύο όψεις του δύο της ίδιας ανησυχίας. Γι' αυτό και θέλω να σας ζητήσω να είσαστε πολύ καθαρός για τις συζητήσεις που γίνονται τώρα για την επιλογή ανάμεσα στην ασφάλεια και το απόρριτο προκειμένου να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Είναι πολύ δικέ οι συζητήσεις που γίνονται. Λοιπόν, υπάρχει κάποια πρακτική τεχνολογική λύση Ευχαριστώ πολύ επίσης τον κύριο Δακίστο για την σε βάθος ανάλυση που κάνει του κειμένου. Δεν θα ρωτήσω, φαντάζομαι ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά. Αυτά που είπατε για την ευθύνη, την υπευθυνότητα, συμφωνούμε πάρα πολύ. Εσείς έχετε την εμπειρία Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε για το επίπεδο στο οποίο χρειάζεται, αλλά εκεί ναι, είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τα μονοπόλια. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ερώτηση και προς εσάς και προς τον κύριο Μπέλτρα και τον κύριο από το Facebook. Το θέμα των μονοπωλίων. Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα του μονοπωλίου γιατί τελικά καταλήγουμε στο καταναλωτές να μην έχουν καμία ελεύθερη επιλογή. Δεν μπορεί να λυθεί από εμά αυτό το θέμα της προστασίας του ιδιωτικού βίου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πρέπει να υπάρχει μια επιπλέον προσήγηση. Πώς θα λυθεί λοιπόν το θέμα αυτό του δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο τελικά μονοπολείται από τη μία πλευρά μόνο. Βλέπουμε όλες αυτές τις ιστορίες στο διαδίκτυο των πραγμάτων που λέμε. Δεν μπορούμε όλα να τα λύσουμε, αλλά σε αυτό το πλαίσιο χάρηκα που άκουσα να λέτε αυτό που τονίζουμε κι εμείς, ότι πρέπει να αποτελεί και μια όθηση στην καινοτομία. Δεν είναι μόνο εμπόδιο, είναι και όθηση στην καινοτομία. Δεν ξέρω. τι άλλες τεχνολογικές λύσεις μπορεί να υπάρξουν. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τις ιδέες σας και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μίκα, ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμες για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ επίσης που θέτετε το θέμα της ασφάλειας. Είναι ένα από τα στοιχεία κλειδί. Και συμφωνώ με την παρατήρησή σας ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συνολική εικόνα, πληροφορίες, δεδομένα, αυτό είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ασφάλεια των δεδομένων, δίκτυα, έχουμε την οδηγία για την ασφάλεια, εντοπισμός και διάδραση. Όταν αρχίζουμε το έργο για τη διάδραση, εσείς αναφερθήκατε στο διαδίκτυο των πραγμάτων και σε μία από τις διαφάνειες είδα κάτι για τη σχέση ανάμεσα στο μηχάνημα και τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλες σχέσεις. Μηχάνημα σε μηχάνημα, σε άνθρωπο σε μηχάνημα κλπ. Μια πολύ πιο περίπλοκη αλυσίδα πραγμάτων. Και τη ισχύει αυτό στην διάδραση δεν είναι όπως ήταν στο Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένου που είχε να κάνει με τον καταναλωτή, το άτομο, τον πελάτη από τη μία και την επιχείρηση από την άλλη και τι γίνεται με την προστασία των δεδομένων και του ιδιωτικού βίου, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις επιπλέον διαστάσεις των σχέσεων. Και ήταν πολύ καλό το παράδειγμα του Facebook. Είναι μια νέα δυνατότητα, μια νέα λειτουργία που προσφέρεται στον κόσμο. Εγώ θέλω να έχω επεξηγήσεις κατά πόσο θα σκοτώσουμε τελικά τέτοιου είδους λύσεις σε αυτή την εκδοχή του κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Θα βάλουμε κάποια ερωτηματικά ή θα βρούμε μια λύση ώστε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδους λειτουργίες θα είναι εφικτές χάρη σε αποφάσεις που θα παίρνουν τα άτομα, γιατί πρέπει να έχουν τον μηχανισμό στη διάθεσή τους να ελέγχουν το τι γίνεται, με τις ρυθμίσεις δηλαδή. Να υπάρξουν νέες δυνατότητες ρυθμίσεων προς τους χρήστες, τους καταναλωτές. Πάντα στον κύριο Τεκίστο γιατί εσείς εκπροσωπείτε την αρχή της προστασίας δεδομένων της χώρας σας. Το πρόβλημα είναι, είμαστε έτοιμοι για εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ελπίζω πως ναι. Συγχρόνως όμως πρέπει να οργανώσουμε τους πόρους μας και τις δυνατότητές μας για να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στον κανονισμό για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό αυτό στα τέλη του 2018. Εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προσπαθούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση το φθινόπωρο με τους εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να δούμε τι κάνουν αυτοί όσον αφορά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί. Για να επανέλθω στους ομιλητές, Ντανιέλ. Ακούσαμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσφορά του κ. Ντεκουίστου. Πολύ δύσκολο βουλευτή να πει τηλεόραση. Μπορεί να θετήσω την προσφορά σα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση ήταν αν αυτός ο κανονισμός ε, θα μας βοηθούσε να βελτιώσουμε την κυβερνοασφάλεια. Όμως ε, νομίζω πρέπει να δούμε με σαφήνεια το άρθρο 6. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω για να βοηθήσουμε σε αυτό γιατί μιλήσατε για το δίκτυο των πραγμάτων, ε, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, όλα αυτά θα γίνουν πολύ πιο σημαντικά ε, όταν θα ισχύει αυτός ο κανονισμός. Και για τα cookies, νομίζω ότι αναφέρθηκε από κάποιους ομιλητές, είμαστε στην εξή κατάσταση. Αν ε, ξέρεις τι είναι ένα cookie, ξέρεις πώς να το βγάλει και από το σύστημά σου. Και αν δεν ξέρεις τι είναι, απλώς κάνεις κλικ και το δέχεσαι. Γιατί θες να μπει στην υπηρεσία που επιθυμείς, θα αλλάξει κάτι, ακόμη και αν θα έχουμε το σύστημα συνένεσης, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι τα κούκκες απλώς ε, θα μπαίνουν γιατί θα θέλουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Έχω και μια ερώτηση, νομίζω αναφέρθηκε το θέμα των υπηρεσιών παρακολούθησης και εντοπισμού. Θέλω να ακούσω την άποψή σας ε, για τις υπηρεσίες video streaming αυτή τη στιγμή. Ε, κάποιες ε, ζητούν ε, εσύ να βάλεις τις υπηρεσίες εντοπισμού στο δικό σου τάμπλετ για να μπορείς να δεις ότι είσαι στην επικράτη που πρέπει να είσαι για να απολαύσεις του δικαιώματο αυτού. Αυτό το κάνουν για να είναι σίγουροι ότι συνάδουν με άλλη νομοθεσία. Και αυτό είναι ένα μεγαλύτερο θέμα, γιατί έχουμε εδώ αντικρούμενη νομοθεσία, έχουμε την οδηγία ψηφιακού περιεχομένου που ε, συζητούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν υπάρχει υποχρέωση στην πρόταση να προσωπηθούν όλα τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα για να μπορούν να επιστραφούν πίσω στον καταναλωτή όταν θα έχουν, ε, θα έχουν τελειώσει οι υπηρεσίε. Ε, τώρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, αναμένεσαι να διατηρεί ανώνυμα τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα για το πώ θα αλληλεπιδρούν όλα αυτά. Και Έχω και μια ερώτηση σε σχέση με το απόρριτο, γιατί βλέπουμε υπηρεσίες όπως το WhatsApp που έχουν κρυπτογράφηση ε, end-to-end από τον ένα χρήστη στον άλλο και πάρα πολύ χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες γιατί είναι κρυπτογραφημένες ε, και ε, αυτό το έκαναν χωρίς κανένα νομικό πλαίσιο, αλλά επειδή το ζήτησε η αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη νομοθεσία σε αυτό. Και σε ό,τι αφορά τώρα βλέπετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την τρομοκρατία και μετά τις επιθέσεις στο Λονδίνο για τις πληροφορίες που υπήρχαν στο WhatsApp νομίζω σε αυτή την περίπτωση. Οι ιδιοκτικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να πάρουν αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει πρόσβαση των διοκτικών αρχών σε τέτοιες υποθέσεις όπου οι πληροφορίες ε, ουσιαστικά κρύβονται μέσω κρυπτογράφησης. Μπορούμε να έχουμε κάποια αναγνώριση αυτού του θέματος στην πρόταση. Ο κύριος ε, Χαντζός, παρακαλώ. Λοιπόν, ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις, αν και νομίζω ότι υπάρχουν διασταυρούμενα σημεία, διασταυρούμενες αναφορές. Να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση για την τρομοκρατία και το απόρριτο έναντι τη σωματικής ασφάλειας, ε, που νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έθεσαν κάποιοι βουλευτές. Να σας, περιγράψω τη δική μας τυχή, τη Semantic. Νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, δεν υπάρχει κάτι απαραίτητα όπως μόνο καλό ή μόνο κακό. Να σας δώσω δύο παραδείγματα συγκεκριμένα μιλάμε, παίρνουμε το χάρη για τη συνένεση ως ε, κάτι καλό. Ε, και είναι καλό να μπορούμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στο χρήστη. Όμω αν εγώ είμαι σε ε, αν το χάρη μπορώ να βάλω ε, ένα παράθυρο που να λέει δέχεσαι αυτό το κούκι, βάλε ε, εντάξει και τότε να κατεβάσει ο χρήστη το μηχανήμα του έναν ιό, Χωρί να το ξέρει. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για κρυπτογράφηση, κρυπτογράφηση είναι μία ε, τεχνολογία ε, βασική και χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο για να προστατεύσουμε τις επικοινωνίες μας, όμως χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση και για να επιτεθεί κάποιος εναντίον μας, παραδείγματος χάρη αν έχει κάποιο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο ουσιαστικά κωδικοποιεί το περιεχόμενο του υπολογιστή σου και κατόπιν οι κακοί ε, σου εκβιάζουν και σου ζητούν χρήματα γι' αυτό. Αναφέρατε και τους τρομοκράτες που χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση ως εργαλείο. Έτσι λοιπόν, είναι ουσιαστικά σαν το μαχαίρι. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να κόψει το ψωμί είτε για να κάνει φόνο. Από τη δική μας σκοπιά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ε, σε ό,τι αφορά την συνεργασία σεβόμενη τις υποχρεώσεις του απερίτου και της ιδιωτικότητας. Εμείς ως βιομηχανία μπορώ να σας πω ότι το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά, είμαστε πολύ διαφανείς για τη συνεργασία που έχουμε με τις διοκτικές αρχές. Εγώ είμαι και ε, στο συμβουλευτικό ε, όργανο της Europol και από την άλλη μπορώ να σας πω ότι θέλουμε να δούμε ποια είναι τα ακριβώς ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Είναι οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και η ευρύτερη ε, συνεργασία ε, σε σχέση με την κρυπτογράφηση. Εμείς συμμετείχαμε σε αυτές τις ζητήσεις, συμμετέχει και η μα μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Όμως ε, θέλω να σας απευθύνω έκκληση προς μια προσέγγιση, δηλαδή ε, ότι θα πρέπει να ε, μην δώσουμε παραδείγματο χάρη ε, πρόσβαση στις διοκτικές αρχές, γιατί παραδείγματος χάρη αν σπάσει κάποιος ε, την κρυπτογράφηση, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον μας. Υπάρχει λοιπόν η πρόκληση για το πώς ακριβώς θα οικοδομήσουμε τη δέουσα διαδικασία για να δώσουμε την πρόσβαση και να είναι δυνατόν να προστατεύουμε τις κοινωνίες μας αλλά και τις τεχνολογίες μας πιο αποτελεσματικά. Κύριε Μπόνι, αναφερθήκατε στην επικοινωνία μεταξύ μηχανών ή ανθρώπου μηχανής και αυτό πρέπει να καλύπτεται στην e-privacy. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας είναι θετικό ότι η Κομισιόν έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή και καλύπτει και τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα. Είναι ουσιαστικό η πρόσβαση στο τελικό σημείο να επιτρέπεται για λόγους ασφαλεία εντός ε, του κανονισμού privacy και να πω ότι είναι ζωτικό και η πρόσβαση για σκοπούς ασφαλείας ε, να μην ε, περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα που καλύπτεται το γενικό κανονισμό κάποιες αντιδράσεις για κάποιες από τις ερωτήσεις σε κάποια που είπε η κυρία Λόριστη Με μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία είδαμε ότι αυτό που αναφέρατε ως ε, μονοπόλιο των δεδομένων, αυτό δεν ισχύει μόνο για το Facebook, αλλά ίσως και για άλλες μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες. Όπως είπατε, δεν θα το λύσει αυτό ο κανονισμός η privacy, αλλά χρειαζόμαστε κάποιες άλλες λύσεις που να λειτουργούν, χάρη και ε, η, επιβολή του νόμου για τον ανταγωνισμό, ε, η επιβολή των καταναλωτικών δικαιωμάτων και ο κανονισμός η privacy. Όμως ε, εδώ θα πρέπει να δούμε αν τελικά ο νικητής θα τα πάρει όλα και αν τελικά το μονοπόλιο θα υπερισχύσει. Αυτό το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τώρα, κινούμαστε προς ένα πιο πολύπλοκο σενάριο, σε έναν κόσμο που οι επικοινωνίες μεταξύ ανθρώπων και μηχανών ε, ε ουσιαστικά θα ε, αλληλεπιδρούν. Μπορούμε να έχουμε και επικοινωνία μηχανής με μηχανή, όμως θέτουμε δύο πολύ βασικές αρχές. Όταν υπάρχει μια υπηρεσία επικοινωνιών μεταξύ μηχανών ή ανθρώπων, θα πρέπει να σέβονται την αρχή του απορρίτου και την αρχή της ασφάλειας. Είπατε ότι τι γίνεται αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ διάφορων δημοσίων συμφερόντων. Παραδείγματο χάρη, η ανάπτυξη των υπηρεσιών θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση εκεί. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν υπάρχει τέτοια σύγκρουση θα πρέπει να δούμε ποιο δημόσιο συμφέρον πρέπει να υπερισχύσει και φυσικά θα πρέπει να μας καθοδηγεί και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για τα όσα είπε κ. Ντάλτον, για το πώς ε, θα βελτιώσουμε την ασφάλεια Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε σωστό ε, πεδίο εφαρμογή αυτών των δύο νομοθετημάτων και να ξανατονίσω τα όσο είπα για τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ζωτικό εδώ. Για την ερώτησή σα για τα cookies, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα τα cookies δεν είναι η κύρια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι του οποίου δεν γνωρίζουν οι καταναλωτέ και ίσω να μην καλύπτονται από την νομοθεσία και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τακίστο, ε, πολύ σύντομα, ε, ορισμένα σημεία. Ε, αρχικά, Συμφωνώ ότι αρκετά από τα σημεία τα οποία, στα οποία αναφέρθηκα χρειάζονται περισσότερο χρόνο και το, η ομάδα εργασίας δημοσίευσε την έκθεση της προσφάτως όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και πρακτικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερα στην ομιλία μου. Ε, και ε, τώρα θα ήθελα ε, να περάσω στα σχόλια του κύριου Μπόνη σχετικά με το πώς προετοιμαζόμαστε για τον επερχόμενο κανονισμό. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η ε, τεχνολογία ε, θα ε, αποτελέσει σημαντικό ρόλο στην απόφαση που θα λάβουμε. Θα ήθελα να αναφέρω την εμπειρία που τον τελευταίο χρόνο όπου το Google είχε μεγάλη δραστηριότητα και πολλές αρχές προσδεδομένων επικεντρώθηκαν πάνω σε αυτό το ζήτημα στο Google και ε, καταφέραμε λοιπόν να προσθέσουμε λύσεις ε, που ε, προσφέρουν προστασία και είμαστε εγκύτερα στους πολίτες. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε τεχνολογίες διότι αν δεν έχουμε την ικανότητα να ε, δουλέψουμε με τις τεχνολογίες τότε υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουμε ένα νέο ψηφιακό χάσμα μεταξύ των αρχών και της εφαρμογής τους. Ε, ο κίνδυνο λοιπόν είναι ότι σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε πώ συγκεκριμένα να εφαρμόσουμε λύσει, τότε ίσω να βρεθούμε σε μια θέση θέση όπου θα έχουμε τις αρχές όμως δεν θα τις εφαρμόζουμε και μακροπρόθεσμα όλο αυτό μπορεί να ε, δημιουργήσει ε, συνέπειες ε, που δεν τις θέλαμε αλλά συνέβησαν. Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια, ε, αναφερθήκατε στην επικοινωνία μεταξύ ε, μηχανών και ανθρώπων ή ε, από μηχανή σε μηχανή σε άνθρωπο. Όσον αφορά την ασφάλεια, εδώ θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή από την πλευρά της, του κανονισμού και εδώ κινούνται από κοινού η ασφάλεια και η ιδιωτική σφαίρα. Δεν είναι πάντοτε ε, αυτός ο κανόνας. Το θέμα είναι η ποιότητα των δεδομένων που είναι ο πυλώνας αυτής της αρχής. Ε, το εργαλείο λοιπόν το οποίο μπορεί να παράσχει την ασφάλεια είναι ε, το ίδιο ε, με αυτά που χρησιμοποιήσουμε ως τώρα, όπως η πολλαπλή ταυτοποίηση ή η, η αποκρυπτογράφηση όλα αυτά ε, προστατεύουν την ιδιωτική ε, ζωή και νομίζω ότι είναι ένα καλό ε, σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Στάς. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε σχετικά με το αν το Facebook ήταν δημόσιο, ιδιωτικό ή όχι και πώς περιλαμβάνεται στο εύρος αυτού του κανονισμού. Ως μηχανικός διστάζω ε, να πω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι. Το Messenger έχει ε, αρκετές ε, ομοιότητες με άλλους Messenger παρόλο που δεν είναι κομμάτι του συνολικού Facebook και επίσης υπάρχει άλλο ένα ερώτημα σχετικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και αυτό υπάγεται ε, στην ομπρέλα της ασφάλειας ε, όπου έχουμε να κάνουμε για την ασφάλεια του πάροχου, του ε, χρήστη. Ε, έτσι λοιπόν δεν θα, αποκλειστούν, ε, μονάχα, δεν αποκλειστεί μονάχα η τρομοκρατία, αλλά ε, εικόνες που χρησιμοποιούνται ε, για απειλή όπως είναι η διοικητική πορνογραφία. Όλα αυτά είναι ένας σημαντικός κίνδυνος ασφάλειας που συμπεριλαμβάνεται σε όλα αυτά. Ο κύριος Μπόνι είχε ένα πολύ καλό ερώτημα εάν όλο αυτό αυτόματα, ε, εάν αυτό θα σκοτώσει το ε, κείμενο το οποίο είδαμε στο βίντεο. Είναι δύσκολο να το ε, πούμε αυτό. Αρχικά θα πρέπει να επεξεργαστούμε τις επικοινωνίες και τα μέσα και δεν γνωρίζουμε το πώς θα λάβουμε την έγκριση από όλους όσοι βλέπουν τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όμως κάνοντας ένα βήμα πίσω ως ε, ε, μηχανικός, όχι του Facebook. Η ανησυχία μου είναι ότι εταιρείε όπως είναι το Facebook θα έχουν ε, δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να καινοτομούν και να αναπτύσσουν τέτοιες τεχνολογίες οι οποίες θα είναι αποκλεισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οι μηχανικοί εντός της Ένωσης δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα είναι αποκλεισμένοι από ολόκληρε αγορές και νέους τομείς που πραγματικά είναι δραστήριοι σήμερα και αυτό είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί, διότι θα πρέπει όλοι να έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν με ένα δίκαιο τρόπο. Ένα ακόμα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το ερώτημα του κ. Ντέλτον για την αποκρυπτογράφηση. Όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια βιώσιμη αγορά όπου οι ε, χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν επιπλέον λειτουργίες ή όχι. Έτσι λοιπόν ε, το ε, Facebook Messenger έχει ένα κρυπτογραφικό κρυπτογραφημένο ε, πλαίσιο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν όμως θα πρέπει ε, να ε, χάσουν ορισμένες λειτουργίες για να μπορέσουμε να έχουμε εμείς πρόσβαση σε αυτό. Μπορούν λοιπόν σε περίπτωση που δεν το θέλουν αυτό να χρησιμοποιήσουν τη μη κρυπτογραφημένη δυνατότητα και μπορούν έτσι λοιπόν να επιλέξουν σχετικά με το ποιο προτιμούν από τα δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στραμ. Έτσι φτάνουμε στο τέλος της ακρόασης αυτής. Βέβαια καμία ακρόαση δεν μπορεί να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι και η συγγήτρια και οι σκιώδες συγγητές νομίζω ότι πιστεύουν πως απαντήθηκαν παρόλα αυτά πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα η συγγήτρια, παρακαλώ τις παρατηρήσεις της, η κυρία Μάριουλα Ορεστίν, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους παρόντες. Έχω μια παρατήρηση. Σε όλη αυτή τη συζήτηση για την ανάγκη που υπάρχει για την προστασία, για το απόρριτο, δεν αναφέραμε όμως κάτι πολύ σημαντικό και αυτό είναι τα παιδιά. Γιατί μπορούμε να μιλάμε, να ξαναμιλάμε για την ε, συνένεση, τη συμφωνία. Τα παιδιά όμως που πριν καλά-καλά αρχίσουν να περπατάνε, αρχίζουν να πιάνουν στα χέρια τους τα smartphones, τα κινητά και τις ταμπλέτες, δεν μπορούμε να μιλάμε για συνένεση από την πλευρά τους πρέπει ορισμού να υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την περίπτωση. Και αυτή είναι νομίζω μια τεράστια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι ευάλωτα και τα οποία χρησιμοποιούν τις ε, έξυπνες αυτές τεχνολογίες χωρίς να είναι σε θέση να προβληματιστούν και να καταλάβουν όλα αυτά τα περίπλοκα νομικά ζητήματα έχουμε να κάνουμε, όπως και αυτοί που φτιάχνουν τα softwares, οι δικηγόροι, οι νομικοί κλπ. Έτσι και εμείς πρέπει να αναγνωρίσουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή είναι λοιπόν η μία μου παρατήρηση. Δεύτερον, τι βγήκε από τη συζήτηση. Βγήκε ότι η εμπιστοσύνη είναι το κύριο στοιχείο για όλους αυτούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες, και για να υπάρχει εμπιστοσύνη πρέπει να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Χρειάζεται διαφάνεια από τη μία και από την άλλη μεριά χρειάζεται διαπαιδαγώγηση του κόσμου. Μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Μπόνι, θέλω και εγώ να έρθω στο θέμα της εφαρμογής των κανόνων. Εντάξει, εγώ είμαι βέβαια καθημαϊκός ε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο μου Ήμουν μαζί με άλλους επόπτες δεδομένων και συναντηθήκαμε με πανεπιστημιακούς και εκεί τέθηκε το ερώτημα ποιος είναι αυτός που καταρτίζει αυτούς οι οποίοι θα γίνουν επόπτες δεδομένων και που θα φροντίσουν και την εφαρμογή όλων αυτών των κανόνων σε όλες αυτές τις οργανώσεις που πρέπει να το κάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα το σωστό προφίλ, γιατί χρειάζεται συνδυασμός γνώσεων, νομικών, πληροφορικής, ε, κοινωνιολογίας και δεν ξέρω τι άλλο. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ναι, υπάρχει το τεχνολογικό ζήτημα, αλλά υπάρχει και το θέμα των ανθρώπινων πόρων. Καμία τεχνολογία δεν μπορεί να τα κάνει όλα από μόνη της. Ωραία, πολλά μας είπατε και μας βοηθήσατε να μάθουμε περισσότερα. Ενισχύσατε τις γνώσεις μας. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εύχομαι στην εισηγήτρια και τους σκιώδες εισηγητές ό,τι καλύτερο για αυτό το ζήτημα. Κάποιοι έχουν φύγει βέβαια. Σας ευχαριστώ πάντως όλους που ήσασταν εδώ, τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν ειδικά για την ακρόαση αυτή. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, λοιπόν, και είμαστε ευγνώμονες.